Καλημέρα σας. Ας, ξεκινήσουμε, οπότε σας παρακαλώ να καθίσετε. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως για τη σημερινή συνεδρίαση. Όπως είχαμε συμφωνήσει εχθές, είχαμε πει ότι θα χρειαστεί ε, το ερωτηματολόγιο με τις πέντε προτεραιότητες σχετικά με τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρακαλούσα μέχρι τις 6 Νοεμβρίου να έχουμε βρει μια συμβιβαστική εναλλακτική σχετικά με την, ε, το ελεγκτικό συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι ένα θέμα όπου θα παρακαλούσα ε, τους ε, υπαλλήλους και τους ευρωβουλευτές να έχουν βρει μέχρι αύριο το πρωί μία λύση για να μπορέσουμε να συντονιστούμε διότι δεν έχουμε πλέον χρόνο. Θέλετε κάτι να πείτε κύριε η κυρία Γκρέσλε και εγώ συζητήσαμε το θέμα για την πολιτική μας ομάδα, δηλαδή η ομάδα του ΕΛΚ ψήφισε ε, χθε έναν συμβιβασμό, τον οποίο ε, είχαμε παραθέσει η κυρία Γκρέσλε και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά ε, βλέπω ότι η μεθοδολογία η οποία έχει επιλεγεί από το Κοινοβούλιο δεν μας ικανοποιεί και δεν έχουμε παρά μόνο μία λύση ε, να ακολουθήσει κανείς ε, το δρόμο του αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο ε, εργάζεται αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημειώνω. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή 2007 διότι όπως θυμάστε παρουσιάστηκε εχθές από τον ε, εισηγητή τον κύριο Σόντεργαντ. Έχετε τον ε, κατάλογο της ψηφοφορίας και υπάρχει απλώς μία προσθήκη στην ε, πρώτη ε, ε, τροπολογία η οποία υπάρχει στο παράρτημα και εάν, εάν δεν έχετε αντίρρηση θα το θα προβούμε εις την ε, ε, στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή για, ε, για το οικονομικό έτος 2007 σχετικά με το Συμβούλιο. Καταρχήν παρά, τροπολογία 14 της κυρίας Αντερέασεν. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας Αντρέασεν Κατά. Η τροπολογία απορρίπτεται. Το δεύτερο θέμα ε, καταπίπτει ε, διότι είναι σχετικό με το προηγούμενο και περνάμε τώρα στην πρόταση του ψηφίσματος σχετικά με την ε, έκθεση. Λοιπόν, καταρχήν τροπολογία 1 η οποία και πάλι έχει υποβληθεί από την κυρία Αντρεάσεν. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Η τροπολογία νούμερο 1 απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 2 που πάντοτε έχει υποβληθεί από την κυρία Αντρέασεν. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 2. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. 2, τροπολογία 3 της κυρίας Γκρέσλε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Πάντα της κυρίας Γκρέσλε. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 ε, του κυρίου Οντί, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην προφορική συμβιβαστική τροπολογία 1 όπως, τροπολογήθηκε, ε, όπως τροποποιήθηκε χθες, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές περνάμε εις ε, την τροπολογία 2 ε, ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται τελική ε, τελική ψηφοφορία με, στην τροποποιημένη έκθεση υπέρ κατά εγκρίνεται μόνο μία διευκρίνηση την οποία μου επισημαίνει η γραμματεία. Πρέπει να ψηφίσουμε επίσης στην αρχή μετά τις δύο τροπολογίες Σεν, δηλαδή την τροπολογία των 14 ε, και 13 πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση ε, για απόφαση στο σύνολό της την πρόταση. Δεν ξέρουμε γιατί μιλάτε. Μπορείτε σας παρακαλώ να το διευκρινίσετε. Μου λέγει η γραμματεία ότι όπως αναγράφεται στον κατάλογο της ψηφοφορίας μετά από την τροπολογία 14 και 13 που παρουσιάστηκαν από την κυρία Αντρέασεν πρέπει να γίνει επιπλέον μία ψηφοφορία επί της πρότασης όπως έχει διατυπωθεί από την κυρία Αντρέασεν. Ε, ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο στη συνέχεια υιοθετήσαμε, υπερψηφίσαμε. Δεν είναι σαφές. Κύριε Πρόεδρε, για να διευκρινίσουμε, πέραν της πρότασης για το ψήφισμα θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, και την απόφαση. Και πρέπει να μετρήσουμε τις ψήφους διότι αυτές θα εγγραφούν στην ε, εγκεκριμένη έκθεση. Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από την τροπολογία 13 γιατί λέγεται ότι η τροπολογία 13 καταπίπτει εάν έχει απορριφθεί το 14. Ουσιαστικά δηλαδή απλούστατα ψηφίζουμε υπέρ ή κατά της ε, απαλλαγής που είναι ένα διαφορετικό θέμα για να ξέρουμε και να μην συγχαίουμε τα πράγματα ουσιαστικά η τελική ψηφοφορία συμπεριλαμβάνει και την ψηφοφορία αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να ψηφίσουμε για να είμαστε πιο σίγουροι, μπορούμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε το, την πρόταση για απόφαση στο σύνολό της αφού απερίφθησαν οι τροπολογίες εν υπέρ κατά Πρέπει να μετρήσουμε παρακαλώ πώς είναι υπέρ και πώς είναι κατά. Κρατήστε τα χέρια σας ψηλά. Κατά. Κατά. Αποχές καμία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Σόντεργαρντ για την εργασία την οποία έκανε και ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα της σημερινής ημερησίας διατάξεως. σχετικά με την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών θα σας αναφέρω τι έγινε χθε στη συνεδρίαση στις 3 μεταξύ του Προέδρου και των συντονιστών των ομάδων διότι θέλαμε απλούστατα να εγκρίνουμε τους εισηγητές των διαφόρων διαδικασιών απαλλαγής για το 2008 και πριν. Ε, πριν το για το 2008 έχουμε τον Λιμπεράσχη για την Επιτροπή. Ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Ματή. Ε, επίσης ε, αποφασίσαμε για τις αποστολές το 2010. Μία αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ελλάδα 27 με 30 Απριλίου, στην Κρατία 1 με 4 Ιουνίου και ε, στην ε, Κροατία 28 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου και τέλος Οκτωβρίου στην Ιταλία. Ε, θα πρέπει οι αντιπροσωπείες να μας κοινοποιήσουν τα 25 μέλη τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτές τις αντιπροσωπείες το ταχύτερο δυνατόν. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε επίσης ε, ε, και ε, να σταθμίσουμε πώς θα κατανεμηθούν οι εργασίες στις ομάδες. Τώρα, ακροάσεις για το 2010. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ε, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις και την νομοθετική εργασία του Συμβουλίου, την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της ε, κοινότητας, διαρθρωτικά ταμεία και αποδέκτες και αναθεώρηση του κανονισμού τέσσερις δηλαδή συνολικά διοργανώσεις για το 2010 και έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες ε, για Απρίλιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο και ε, θα πρέπει επιγόντως ε, να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τις ε, μελέτες του 2009 σχετικά με τα συστήματα διαχειρίσεως του, των διαστορτικών ταμείων όπου είναι εισηγητής ο κύριος Λιμπεράτσκι και το ΕΛΚ θα μας κοινοποιήσει για το, τη δεύτερη έκθεση και θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε ε, και άλλα θέματα τα οποία έχουμε κάπως προγραμματίσει χωρίς όμως να έχουμε αποφασίσει τελεσίδικα διότι αυτό θα γίνει το 2010. Στη συνέχεια προβλέψαμε μία ακρόαση για τους νέους επιτρόπους, ε, είτε νέους είτε αυτούς των οποίων η θητεία θα ανανεωθεί και ακολουθήσαμε ε, τις, ε, ε, τις υποδείξεις της διασκέψεως των Προέδρων 25-26 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και από τις 30 μέχρι τις 4 στις Βρυξέλλες. Δηλαδή η διάσκεψη των Προέδρων παρουσίασε ένα πολύ εκτενές ε, ε, ερωτηματολόγιο που θα απευθυνθεί σε όλους τους ε, επιτρόπου, υποψηφίους επιτρόπους αλλά η Επιτροπή μας ήθελε να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις ιδίως όσον αφορά την, τα συγκεκριμένα θέματα. Οπότε περιμένουμε να έχουμε, να έχουμε συντάξει το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα υποβάλουμε εις τους συντονιστές και έχουμε επίσης στους επιτρόπους και έχουμε για τους συντονιστές ορισμένα θέματα για το ελεγκτικό συνέδριο. Διότι όπως ξέρετε, εννέα μέλη από το Μάιο έως τον Νοέμβριο, του χρόνου θα λήξει η θητεία τους και πρέπει να διορίσουμε καινούριου με ακροάσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι υποψήφοι για το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε μετά και ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος για τις συνεδριάσεις όλου του 2010 της Επιτροπής μας, ελέγχου του προϋπολογισμού και το πρόγραμμα για την επίσκεψη του ελεγκτικού συνεδρίου σήμερα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να πετύσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο έτσι όπως θα οριστούν και από τις ε, τρεις βασικές πολιτικές ομάδες. Ο διευθυντής της Όλαφ ζήτησε από την Κομισιόν να επισκεφθεί το γραφείο της Όλαφ μας έδωσε ημερομηνίες και δώσαμε εντολή στη γραμματεία για το Μάρτιο όλα αυτά. Τώρα, ορισμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου κάνουν μία απόπειρα να υποκαταστήσουν την Επιτροπή μας του Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και το τελευταίο γεγονός ήταν αυτό με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και εγώ απάντησα ήδη στον πρόεδρο της ε, διάσκεψης των πρόεδρων των Επιτροπών, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ότι δεν υπήρχε επικάλυψη σε ένα θέμα το οποίο είναι θέμα καθαρά της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ζητήσαμε από, τη γραμμα... τις γραμματείες να βρούνε μία λύση. Και είπαμε ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μπορεί κάλλιστα να γνωμοδοτήσει σχετικά, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Τώρα για τα άλλα σημεία, για το πρακτικό της 20 Ιουλίου του 2009 γιατί ο κύριος Αντρίσεν είχε θέσει τότε ένα θέμα για να έχει τα ονόματα των μελών της Επιτροπής ε, και μετά επίσης ε, υπήρχε και ένα θέμα προβλημάτων με την ε, ψηφοφορία που είχαμε καταλήξει να τη βάλουμε στην επόμενη ε, συνεδρίαση για να ψηφιστεί διασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες σε μια πρώτη φάση για την ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα, σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης είναι η ειδική έκθεση 6 κάθετος 2009 του Ελεκτικού Συνεδρίου «Επισητιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άπορους, αξιολόγηση των στόχων, των μέσων και των εφαρμοζομένων μεθόδων». Η η συγγήτρια η κυρία Ντελόνζ έχει το λόγο. Δεν τη βλέπω και αφού δεν τη βλέπω φυσικά δεν μπορεί να μιλήσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Να δώσουμε τον... Περιμένοντας λοιπόν την κυρία Ντελόνγκ, την οποία θα την ψάξουμε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Αλάς, εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι εδώ ο κύριος Αλάς? Εκεί, εκεί. Α. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, στη σύντομη παρουσίασή μου θα σα δώσω μία σύντομη επισκόπηση των βασικών συμπερασμάτων τη εργασία μα για την στη βοήθεια για του απόρου. Το πρόγραμμα εισήχθη ως αντίδραση στις καταστάσεις ε, έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του σκληρού χειμώνα του 1987 όταν η κοινότητα αποφάσισε να δώσει γεωργικά προϊόντα χωρίς ε, τέλη σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για να διανεμηθούν σε άτομα που το χρειάζονται. Το μέτρο λοιπόν αυτό ε, ισχύει ακόμα σήμερα και χαιρετίστηκε από τότε με ενθουσιασμό. Η ένδια αποτελεί ακόμα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, το οποίο χειροτερεύει λόγω τη κρίση. Σύμφωνα με τις στατιστικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρώπη των 27 υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κίνδυνο ένδυα. 53 εκατομμύρια δηλαδή στα κράτη-μέλη. Είναι πολλές χιλιάδες οι οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με την παροχή βοήθειας Ο αριθμός των τελικών δικαιούχων εκτιμάται ότι είναι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι σε τίσεο επίπεδο, αν και κατά μέσο όρο καθένας τους λαμβάνει ένα γεύμα ανά μήνα και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος από 307 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 500 εκατομμύρια ευρώ το 2009. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα είναι θελούσια και ουσιαστικά σήμερα συμμετέχουν 19 κράτη-μέλη. Σε λειτουργικό επίπεδο, στα κράτη-μέλη, το πρόγραμμα το διαχειρίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών. Ο έλεγχος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου εστιάστηκε στο περιεχόμενο της ε, αγοράς η οποία εξελίσσεται και της κοινωνικής ε, κατάστασης και της καταλληλότητας των μέτρων που λαμβάνονται. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τα έξι συμπεράσματα και τις εξή συστάσεις. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο βασικούς στόχους στο πρόγραμμα, δηλαδή αφενός να γίνει μια σημαντική συμβολή για την ευημερία των ε, απόρων και αφετέρου να σταθεροποιηθεί η αγορά των γεωργικών προϊόντων, με την μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης. Ουσιαστικά αυτός ο στόχος ο οποίος κυριαρχεί είναι ο κοινωνικός στόχος και η χρηματοδότηση του προγράμματος από την ε, ΚΑΠ ήταν δικαιολογημένος. Ωστόσο, όπου μειώθηκαν τα αποθέματα παρέμβασης σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο πρόσφατα, στα πρόσφατα χρόνια, η σημαντική μείωση στα αποθέματα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο να αγοράζονται στην αγορά 85% των προϊόντων αυτών για διανομή. Άρα το ελεγκτικό συνέδριο συστήνει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχιστεί η χρηματοδότηση από το ΚΑΠ. Σε γενικές γραμμές ε, δεν υπήρχε επαρκή συντονισμός με άλλους βασικούς φορείς για κοινωνική δράση στα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα και είναι απαραίτητη αυτή η συνεργασία για την καλύτερη κατανόηση του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ε, και να λάβουν κίνητρα προκειμένου να εντάξουν το πρόγραμμα αυτό στο γενικότερο πλαίσιο κοινωνική πολιτική του. Το μέτρο σχεδιάστηκε για να απαλύνει την φτώχεια, όχι όμως για να την εξαλείψει. Ως, εκ τούτου οι πόροι αυτοί έχουν περιορισμένη μόνο αντίκτυπο στην κατάσταση των απόρων. Τους δίνουν δηλαδή κατά μέσο όρο ένα γεύμα το μήνα. Άρα, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, είναι απαραίτητο να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες και να τεθούν οι σωστοί στόχοι. Οι φυσάμενες διατάξεις περιορίζουν την ε, ποικιλία των προϊόντων που διανέμονται, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην όλη των διανομής ε, σημαίνουν ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των τελικών δικαιούχων. Γι' αυτό λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο συστήνει να υπάρξουν ρυθμιστικοί προορισμοί προκειμένου να δοθεί, αν θέλετε, η κατάλληλη η κατάλληλη συμπληρωματικότητα, η κατάλληλη διατροφική αξία των τροφίμων που διανέμονται. Επιπλέον, το συνέδριο εντόπισε κάποιες αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης και πρότεινε και σχετικές λύσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι το, Σεπτέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την βελτίωση, για την τροποποίηση, συγγνώμη, του σχετικού κανονισμού του Συμβουλίου που έγκρινε το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2009. Η πρόταση αυτή αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη διαμόρφωση νέου νομικού πλαισίου για το πρόγραμμα και αν εφαρμοστεί θα λύσει κάποιες από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας κάνατε και την ε, εισαγωγή για θέματα τόσο σημαντικά. Ήρθε και η συγγήτρια, της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη και ενώπιν του συνεδρίου που δεν ήμουν στην ώρα μου. Στην... Έπρεπε να είμαι στην άλλη επιτροπή στην οποία συμμετέχω και ξέρω ότι μιλάμε και για κλωνοποίηση ζώων και ξέρω ότι είναι αμφιλεγόμενο το θέμα αυτό, αλλά μακάρι να μπορούσαμε να κλινοποιήσουμε και του πολιτικού για να είναι σε διάφορε επιτροπέ. Να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την εισαγωγή που έκαναν και τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής σε ό,τι αφορά τη μετάφραση, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό, τη μετάφραση δηλαδή αυτών των συστάσεων σε πρακτικά μέτρα για το μέλλον. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε ε, δύο-τρία συμπεράσματα τα οποία αναφέρονται και στο έγγραφό μου. Το είπε και το συνέδριο, βρισκόμαστε σε μια φάση νομοθεσίας για να τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί το εκτελεστικό πρόγραμμα και είναι πολύ ε, πραγματικά απαραίτητη η προσαρμογή αυτή στην παρούσα φάση για το έγγραφο εργασίας μου σημείωσα ότι τα ερωτηματικά ή παρατηρήσεις τι οποίες θέτει το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την νομοθετική βάση της νομοθετική πρότασης θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σαφήνεια. Γιατί όλα ξεκινάνε φυσικά από την νομική βάση. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι θα ήθελα να τονίσω το εξή, το οποίο επίσης αναφέρω στο έγγραφο εργασίας μας η ανάγκη, η επιστηστική βοήθεια να στοχοθετηθεί καλύτερα, να τεθούν πιο σωστές προτεραιότητες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για όσους πραγματικά τη χρειάζονται. Γιατί αν υπάρχουν πιο σαφή κριτήρια, αν, υπάρχουν, αν υπάρχει πιο σαφή σε προστιθέμενη αξία, νομίζω ότι ε, έτσι αξιοποιείται καλύτερα ε, αξιοποιούνται καλύτερα οι ευρωπαϊκοί πόροι. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο έγγραφο εργασίας μου, καθώς και πολλά άλλα στοιχεία. Ελπίζω ότι το έγγραφο αυτό θα μας συνοδεύσει για την υπόλοιπη νομοθετική διαδικασία, για την διαμόρφωση του νέου προγράμματος, αλλά και σε άλλες στιγμές ενδεχομένως της νομοθετικής μας διαδικασίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ελεκτικό συνέδριο και η συγγήτρια εξήγησαν τις λεπτομέρειες για το υπόβαθρο της πρότασης αυτής που αρχικά ήταν ε, συνδεδεμένο με το ΚΑΠ και με τα γεωργικά προϊόντα που υπήρχε πλεόνασμα και τώρα φαίνεται ότι μειώνεται αυτός ο σύνδεσμος καθώς ε, μειώνονται και τα γεωργικά αποθέματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τα της χρηματοδότησης ε, από την ΚΑΠ. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον του προγράμματος γιατί είπαμε ότι εξατλείται τα αποθέματα και αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Τι θα συνεχίσει να χορηγείται στους δικαιούχους. Ωστόσο, θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε ενδεχόμενη χρηματοδότηση από άλλη γραμμή του προϋπολογισμού. Να βγει από την ΚΑΠ, να τοποθετηθεί σε ξεχωριστή γραμμή. Επίσης, να κοιτάξουμε τα κριτήρια για την ε, κατανομή των πόρων προκειμένου, όπως είπε και η συγκέντρια, να γίνει καλύτερη στοχοθέτηση, καλύτερη θέση προτεραιοτήτων και όλα αυτά να τα δούμε και στην επόμενη διαδικασία απαλλαγή του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ναι, να, να πω στου συναδέλφου ότι κάθε φορά που πηγαίνω στον πατέρα μου στην Κρήτη μα δίνει τρόφιμα από τα αποθέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι λοιπόν από πού προέρχονται. Γιατί μα τα δίνουν έτσι, χωρίς ε, αντάλλαγμα. Έτσι πάει. Μακαρόνια, ε, σκόνη γάλακτος και όλοι μου λένε ότι αυτά είναι από θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει λοιπόν δικαίωμα πατέρα να τα πάρει αυτά τα α, τρόφιμα, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια, πολύ αλλά τέλος πάντων δεν το δικαιούται, αλλά παρόλα αυτά τα λαμβάνει. Γιατί, γιατί τα κριτήρια επιλογής δεν είναι αρκετά σωστά και το λέει και η συγγήτρια στην έκθεσή της ότι τα κριτήρια διανομής δεν επαρκούν. Καταρχάς όμως θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ του προγράμματος γιατί ο πατέρας μου και ο γειτονά του είναι πεπισμένοι ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά φυσικά δεν έχει νόημα να καταλήγουν τα τρόφιμα αυτά σε λάθο ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε σαφή ορισμό, σαφή ορισμού. Και αυτό το απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι ο υπεύθυνο, ποιοι μπορεί να κάνουν τέτοια διανομή. Γιατί να λέμε έτσι απλά φιλανθρωπικές οργανώσεις, ε, δεν αρκεί αυτό. Έχει χρήματα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετάμε αυτό το δύσκολο θέμα στη μέση και δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι η κατάλληλη οργάνωση. Και τελικά τι γίνεται, δεν έχουμε την αποδοτικότητα που θα έπρεπε να έχουμε, την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί και δεδομένη της οικονομικής κρίσης, η οποία είναι έντονα σε αρκετές χώρες, είναι πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια, μην την υποτιμούμε. Απλά θα πρέπει να καταλήγει στα κατάλληλα χέρια. Και επίσης να προσέξουμε, και αυτό το λέω και πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο follow-up να ελεγχθεί όχι αν σωστά έγιναν οι δαπάνες, αλλά αν σωστά, σωστά χέρια κατέληξαν. Ε, κύριε Ντελάνγκε, ναι. Να θέσω μία ερώτηση κατευθείαν κι εγώ. Γιατί κοιτώντα πώ γίνεται η κατανομή των πόρων σήμερα, εντό του σημερινού προγράμματο, σημαντικό τμήμα, αν σωστά κατάλαβα, 70%, 3 τέταρτα περίπου, καταλήγει σε μεγάλα πλούσια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι από μία χώρα η οποία είναι σε σκληρή γραμμή. Λέει ότι αυτή είναι η κοινωνική μα ε, ε, πολιτική και αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτή την ε, σκληρή γραμμή εγώ δεν την ακολουθώ γιατί θεωρώ ότι μια αξιόπιστη αρχή δεν μπορεί να σταματήσει από τη μια μέρα στην άλλη ένα τέτοιο καλό σύστημα. Άρα λέω μέχρι το 2013 να μείνει το σύστημα όσο έχει και μετά να δούμε τι γίνεται και να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς θα είναι στη συνέχεια το πρόγραμμα αυτό και αν θα πάρει μια συνολική ευρωπαϊκή διάσταση. Μέχρι το 2013 όμως το θέμα είναι να γίνει καλύτερη στοχοθέτηση για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το 70-75% των πόρων αυτών να καταλήγει σε μεγάλα κρατημέλη. κράτη-μέλη. Μήπως θα ήταν μια ιδέα να πούμε, κοιτάξτε, ας κρατήσουμε τον προπολογισμό αυτό που έχουμε σήμερα, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά όπως είπε και στον συνάδελφος. Ποιες είναι οι οργανώσει που κάνουν τη διανομή. Δεν είναι δυνατόν τα χρήματα αυτά να ε, ωφελούν σχεδόν αποκλειστικά τις περιοχές εκείνες, τις περιφέρειες εκείνες όπου το ΑΕΠ δεν είναι χαμηλότερο του ευρωπαϊκού όρου. να μην το σταματήσουμε το πρόγραμμα αυτό κατευθείαν, αλλά να το κάνουμε πιο δίκαιο. Θα ήθελα να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα σχόλια. Το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομίσιον σχετικά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και την, κυρία Ντελάνα για την έκθεσή της το έγγραφο εργασίας της μάλλον. Μια ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Το βασικό στοιχείο της έκθεσης είναι ασφαλώς το γεγονός ότι τίθεται ένα αμφιβόλο ο σύνδεσμος του προγράμματος με, τη, με τα έξοδα της ΚΑΠ. Η κοινωνική διάσταση φαίνεται να είναι πιο σημαντική από ότι ε, η δικλίδα για τα αποθέματα τα γεωργικά. Η Κομισιόν διαφωνεί με το αξίωμα αυτό. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο πρόγραμμα, την επιστική ασφάλεια για τους απόρους και κατά δεύτερον μία εναλλακτική ε, διέξοδο για τα αποθέματα ε, παρέμβασης. Και αυτό ορίζεται από το άρθρο 53 της συνθήκης. Και να σας πω ότι για το πρόγραμμα 2009-2010, Πρόεδρε, το οποίο θα αποφασιστεί αυτή την εβδομάδα περίπου το 90% του προπολογισμού των 500 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί μέσω ε, αποθεμάτων παρέμβασης. Άρα φέτος έχουμε επαρκή αποθέματα. Περίπου 90% κύριε Πρόεδρε. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφή αυτό ο σύνδεσμο μετά από θέματα παρέμβαση και όλα αυτά σε ό,τι αφορά 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι 20 είναι τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν φέτο, όχι 19. Έχουμε και ένα κράτο μέλο επιπλέον, το οποίο επέδειξε ενθουσιασμό για το πρόγραμμα. Και φυσικά τίθεται λοιπόν το ερώτημα, καταλήγουν τα τρόφιμα αυτά στους πλέον απόρους της Ευρώπης. Εμείς στις ε, Βρυξέλλες, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι πιο άποροι αυτοί σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε όμως ένα πρώτο κριτήριο για την διανομή, την κατανομή του προϋπολογισμού αν θέλετε και το 2009 εγκρίναμε μια νέα μεθοδολογία η οποία αντικατοπτρίζει με καλύτερο τρόπο τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου για την καλύτερη στοχοθέτηση και χρήση των πόρων. Ε, συνδυάζουμε το κριτήριο του κινδύνου ένδυας με την κατάσταση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Άρα έχουμε ήδη προσαρμόσει τα κριτήρια κατανομής. Και πρόεδρε για να συνεχίσω, ο προϋπολογισμός αυτός στη συνέχεια κατανέμεται στις ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις και φυσικά ε, στηριζόμαστε σε αυτές να καθορίσουν στη συνέχεια ποιοι είναι οι πιο άποροι της Ευρώπης. Στην κατανομή λοιπόν των τροφίμων, το πρόγραμμα μας μεταξύ 30 και 60% συγγνώμη, 30 και 70% ε, αποτελεί την πηγή των τροφίμων που διανέμουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το πρόγραμμά μας για τις ε, οργανώσεις αυτές αν ο κ. Χατζημαρκάκης λέει ότι ο πατέρας του δεν είναι αρκετά φτωχός για να λαμβάνει τέτοιους, ε, τέτοια τρόφιμα, ε, δεν ξέρω τον πατέρα του, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και να απευθυνθεί κανείς στη φιλανθρωπική οργάνωση επιτόπου για να εξετάσει την κατάσταση αυτή. Επί της αρχής όμως, ορίζω οποιαδήποτε πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα η κατανομή μέσω των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Αυτές είναι, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ε, απόρων. Επίσης σημαντικό στο πλαίσιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξή ότι το Κοινοβούλιο με συνέπεια έχει υποστηρίξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το πρόγραμμα αυτό έχει αυξήσει τον προπολογισμό του ακόμα και πέρα από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και την τελευταία φορά που υποβάλαμε πρόταση, κύριε Πρόεδρε, ε, με συντριπτική πλειοψηφία το Κοινοβούλιο, με 425 ψήφους ε, υποστήριξε το Κοινοβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συνεχίσει το πρόγραμμα με αναφερμένο όμω τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν μου προκαλεί κάπω έκπληξη το γεγονό ότι στο έγγραφο εργασία βλέπω να υπάρχουν και να αντιτυπώνονται κάποιε αμφιβολίε για την νομική βάση. Καταρχά, υπήρξε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Συμφώνησε το Κοινοβούλιο με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και την νομική βάση. Και εξ όσων γνωρίζω, Πρόεδρε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν ε, διενέργησε ε, νομική ανάλυση της νομικής αυτής βάσης. Συγγνώμη, ναι, νομική βάση, νομική ανάλυση της νομικής βάσης. Επίσης αναφέρεται, αναφέρονται κάποιες προτάσεις βελτίωσης, αλλά επίσης αναγνωρίζεται ότι η πρότασή μας και η πρόταση του Συμβουλίου αντιμετωπίζει τα βασικά σημεία τα οποία επικρίνει το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή η πρόταση έγινε και πριν από τη δημοσίευση του ελεγκτικού συνεδρίου, μη σας πω. Άρα, στην πρότασή μας, ήδη αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια θέματα. Για να μην περιοριστούν, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις, συγγνώμη, οι διανομές στα αποθέματα παρέμβαση. Άλλα σημεία κριτικής σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ε, για τους διαγωνισμούς και αυτό θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής. Άρα, συνοψίζοντας, Πρόεδρε, το βασικό φυσικά είναι η νομική βάση και εκεί κατανοούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει αυτή την ε, επέκταση, την τροποποίηση στην ίδια νομική βάση και γι' αυτό λίγο μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι βλέπουμε στο έγγραφο εργασία να αμφισβητείται αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελάνε. Δύο απαντήσεις να σας δώσω. Να δώσω στις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, η πρώτη πρόταση των συμπερασμάτων του εγγράφου εργασίας όπου αναφέρεται ότι δεν χαιρετίζουμε μόνο το έλεγχο του συνεδρίου αλλά και την τροποποιημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά να επαναλάβω ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει προβεί σε κάποιες δηλώσεις και σε κάποιες παρατηρήσεις για την νομική βάση. Το ίδιο και αρκετοί συνάδελφοι. Το μόνο που λέμε δηλαδή είναι ότι το παίρνουμε στα σοβαρά το θέμα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη στις συζητήσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν γράφω κάτι που δεν ισχύει. Επίσης να υποδείξω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την προτελευταία, το προτελευταίο μου συμπέρασμα ότι φυσικά σωστό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τις φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες επιτόπου ε, διανέμουν τα τρόφιμα αυτά και αυτό δεν μπορεί να συμβεί φυσικά κεντρικά από τις ε, αλλά κοιτώντα το άρθρο 274. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που παραμένει υπεύθυνη για το τι γίνεται με τα χρήματα αυτά και που καταλήγουν. Άρα, υπό την έννοια αυτή, η έκθεση του συνεδρίου αποτελεί έναν τρόπο για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει και να καταλάβει ποιες είναι οι αρμοδιότητές της βάσει του άρθρου 274. Και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω ε, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας έχει τις δικές του αρμοδιότητες για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους αυτούς. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, πάμε στην επόμενη έκθεση. Η ειδική έκθεση 9 κάθετος 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα και απόδοση των δραστηριοτήτων επιλογής προσωπικού. Πρόκειται για μία σημαντική έκθεση η οποία αποτελεί και αντικείμενο διαφωνίας ε, εντό αγωγικών διαφωνία με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η κυρία Γέντρεγεύσκα έχει το λόγο. μου είπανε ότι θέλετε να ακούσουμε πρώτα τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Η κυρία Ιρένα Πετρούσκεβιτσένε. Συγγνώμη αν δεν το πρόφερα καλά το όνομα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριοι Ευρωβουλευτές, Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να, παρουσιάσουμε ε, την έκθεσή μας για την αποτελεσματικότητα της ΕΠΣΟ αλλά εφόσον υπάρχει το γραπτό μας κείμενο και παρουσιάζει σωστά την ε, ουσία της εκθέσεώς μου καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθώ μόνο σε ορισμένα θέματα οπότε θα είμαι σύντομη στην αρχική μου παρουσίαση και θα απαντήσω σε ό,τι συγκεκριμένες ερωτήσεις έχετε. Καταρχήν θα ήθελα να παρουσιάσω το γενικό πλαίσιο σχετικά με αυτό τον οικονομικό έλεγχο που ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων επιλογής προσωπικού της ΕΠΣΟ. Όπως γνωρίζετε από το 2003 όλες οι ανοιχτές, όλοι οι ανοιχτοί διαγωνισμοί για την επιλογή δυνητικού προσωπικού ε, έχει διοργανωθεί, έχουν διοργανωθεί από την ΕΠΣΟ και ε, ε, με την διεύρυνση υπήρξαν πολύ περισσότερες προσλήψεις και δεν μπορούσε το κάθε θεσμικό ε, όργανο να τις αντιμετωπίσει χωριστά και γι' αυτό και η ΕΠΣΟ από κοινή απόφαση όλων των θεσμικών οργάνων απέκτησε τη δυνατότητα να οργανώνει τις διαδικασίες επιλογής. Είναι ένα διαθεσμικό όργανο και αυτή είναι και η πρώτη ε, ιδιομορφία αυτής, ε, αυτού του ελέγχου διότι ε, διοικητικά η έψο είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δεν ελέγχουμε μόνο την Επιτροπή αλλά και ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΟ που ε, αντιπροσωπεύονται όλα τα θεσμικά όργανα. Το βασικό στόχος ήταν να καθορίσουμε αν ε, οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού της ΕΠΣΟ ήταν αποτελεσματικές. Και εδώ θέλω να πω ότι η ΕΠΣΟ αναλάβει την διαδικασία επιλογής αλλά η ευθύνη για την πρόσληψη παραμένει σε κάθε θεσμικό όργανο. Η ΕΨΟ απλούστατα παρουσιάζει έναν κατάλογο αλλά από τις, τα θεσμικά όργανα εξαρτάται εάν θα προσλάβουν τους επιτυχείς ε, υποψηφίους από τους καταλόγους αυτούς. Ο έλεγχος ε, δεν περιέλαβε την ε, πρόσληψη διότι θα χρειάζεται χρειαζόταν μια διαφορετική, ένας διαφορετικός έλεγχος της πολιτικής προσλήψεως των θεσμικών οργάνων. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε, ένα, σε μια δεύτερη ιδιομορφία του ελέγχου, διότι όταν τελειώσαμε την αρχική μας εργασία ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΟ υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2008 το πρόγραμμα αναπτύξεω της ΕΠΣΟ, EDP, το οποίο ε, ε, επιλύει πολλές πολλές από τις αδυναμίες τις οποίες είχαμε εντοπίσει κατά τον έλεγχο. Οπότε λάβαμε υπόψη ή στον έλεγχό μας το EDP αλλά ε, μόνο σε ό,τι αναφερόταν στα θέματα του ελέγχου μας. <clears throat> Και αυτό το οποίο παρουσιάζουμε στην έκθεσή μας δεν είναι ε, έλεγχος του προγράμματος αυτό του EDP απλούστατα οι συστάσεις μας λαμβάνουν υπόψη αυτά τα οποία προβλέπονται μέσω του EDP σχετικά τώρα με ε, τις, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά μας. Το συμπέρασμα είναι ότι η ΕΠΣΟ κατάφερε επιτυχώς να αυξήσει τον αριθμό των ανοιχτών διαγωνισμών που απαιτήθηκαν από την διεύρυνση. Αλλά υπήρξαν ε, τέσσερα ε, βασικά μειονεκτήματα ε, για την αποτελεσματικότητα της ΕΠΣΟ. Καταρχήν, οι ανάγκες προσωπικού δεν κοινοποιούνται στην ΕΠΣΟ εγκαίρως και δεν βασίζονται σε μία συνεκτική μεθοδολογία. Επιπλέον δεν υπάρχει μία κοινή μέθοδος ε, για να ε, μπορέσουν να αξιολογηθούν οι ανάγκες αυτές από την έψω και τα θεσμικά όργανα. Η έλλειψη λοιπόν των ε, έγκαιρων πληροφοριών από τα θεσμικά όργανα σχετικά με τις ανάγκες προσωπικού και η έλλειψη κοινή μεθοδολογίας οδήγησε σε καθυστερήσεις ή την διαδικασία επιλογής και ε, πολλές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Δεύτερη αδυναμία, η την διαδικασια επιλογης και πολλες αλλαγες στις τελευταίες στιγμης δευτερη αδυναμια η διαδικασια της, επιλογής προσωπικού ήταν πολύ μακριά και σχετικά με τα πρότυπα της ΕΠΣΟ και ακόμη και με την ε, ε, διεθνή βέλτιστη πρακτική ε, Αυτέ αυτές οι διαδικασίες οδήγησαν ότι τα θεσμικά ε, όργανα δεν μπόρεσαν να προσλάβουν τους υποψηφίους όποτε τους χρειαζόντουσαν ε, και μπορεί να απογοητεύσουν και καλούς υποψηφίους από την αρχή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ε, τρίτη έλλειψη ε, μπόρεσαν οι διαγωνισμοί αυτοί ε, να αποδώσουν μόνο δύο τρίτα του αριθμού των επιτυχόντων και ε, δεν καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες του κανονισμού οι οποίες προβλέπουν ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν τουλάχιστον τόσα ονόματα υποψηφίων όσο και οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν και ότι ε, θα πρέπει οι υπάλληλοι να προέρχονται από το ευρύτερο γεωγραφικό πολιτικό φάσμα των κρατών μελών και ε, να καλύψουν τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων δεν μπόρεσε κανείς να θεωρήσει τέταρτη αδυναμία αυτή ότι η πληροφόρηση για τη διαχείριση της ΕΠΣΟ ήταν αξιόπιστη ε, σχετικά με το κόστος της ε, τοποθέτησης ενός επιτυχόντος στον κατάλογο ε, των επιτυχόντων και το πρόγραμμα δεν έχει καμία ένδειξη σχετικά με το δυνητικό κόστος κόστος και τα μελλοντικά ωφέλη από το EDP. Αυτές ήταν ε, οι αδυναμίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από την Δημοσιονομική Αρχή. Τέλος, οι ε, συστάσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο έκανε οκτώ συστάσεις. Η πρώτη και η δεύτερη ε, δεν απευθύνονται στην ΕΠΣΟ, αλλά οι σταθεσμικά όργανα, τα οποία οι εκπρόσωποι ε, συνιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΟ και αναφέρονται εις καλύτερο προγραμματισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής. Δηλαδή, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να δίδουν συνέψω ενγέρο εγκαίρως τις πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες προσωπικού βάσει μιας κοινή μεθόδου για αξιολόγηση των αναγκών και με ένα κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα. Ε, ε, η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής προσωπικού θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη της ότι ε, θα χρειαστεί η στήριξη ε, από επαγγελματίες πολιτικά Συμβούλια Επιλογής για να μπορέσει να επιλεγεί το καλύτερο προσωπικό. Οι συστάσεις 3 έως 6 αναφέρονται στο, στην καλύτερη απόδοση των διαγωνισμών και από πλευράς αριθμών και από πλευράς γεωγραφικής κατανομής. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες γλωσσικές ανάγκες, προεπιλογή είχε γίνει στο παρελθόν μόνο σε τρεις γλώσσες αλλά ε, για να τονίσουμε περισσότερο τις επαγγελματικές παρά τις γλωσσικές δεξιότητες το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά ε, να γίνεται η προεπιλογή και στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, όσον αφορά τις ανακοινώσεις για τους διαγωνισμούς, το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά η ΕΠΣΟ να εφαρμόσει πιο αυστηρά τους μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου για να εξασφαλίσει ότι θα είναι σαφής και ε, μία άλλη σύσταση αναφέρθηκε στον αριθμό ε, των υποψηφίων για κάθε διαδικασία ε, και για κοινή δράση όλων των θεσμικών οργάνων για να αναπτύξουν και να χρηματοδοτήσουν μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας για το συντονισμό της ΕΠΣΟ κατά τρόπον ώστε να καλούνται, καλείται ένας αριθμός επαρκής υποψηφίων για περαιτέρω εξετάσεις. Ε, τέλος, όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία, συνιστούμε ε, η ΕΠΣΟ να αναλύσει τις λόγους των γεωγραφικών ε, ανισορροπιών και να προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα. Τέλος, αναφέρομαι σε δύο συστάσεις που αναφέρονται στην πληροφόρηση από πλευράς της διοίκησης το, και για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το κόστος των διαγωνισμών η ΕΠΣΟ θα πρέπει να εντοπίσει το κόστος του προϋπολογισμού για να τοποθετηθεί ένας υποψήφιος στον κατάλογο των ε, ε, επιτυχόντων και ε, να μπορέσει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα EDP για να διευκολυθεί η ε, λειτουργία της δημοσιονομικής αρχής και η χρηματοδότηση του προγράμματος για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους διαγωνισμούς του χρόνου το ελεκτικό συνέδριο συνιστά η ΕΠΣΟ να αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες δηλαδή να εξασφαλίσει ότι η Τράπεζα Δεδομένων θα αποφύγει ε, την ε, παρίσφρηση ε, πολλαπλών υποψηφιωτήτων ότι θα χρησιμοποιηθεί ε, συνεκτικά σε όλους τους διαγωνισμούς και ότι θα επιτρέψει να υπάρξουν έγκαιρες σωστές πληροφορίες διοικητικές και στο επίπεδο του διαγωνισμού και γενικότερα. Γενικώ όμως πιστεύουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη στήριξη των θεσμικών οργάνων, δηλαδή θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να δίνουν εν εγκαίρως τις πληροφορίες στην ΕΠΣΟ, ιδίω όσον αφορά τον ε, τριετή μελλοντικό προγραμματισμό και ε, για να υπάρχουν ε, επαρκείς ειδικευμένοι αξιολογητές στην ΕΠΣΟ. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα θελήσετε να μου υποβάλλετε. Η κυρία Γεντρογεϊεύσκα, η συγγήτρια. Ε, dziękuję panie przewodniczący. Będę I speak θα μιλήσω στα αγγλικά νομίζω για να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα. Και επίσης επειδή έγραψα το έγγραφο εργασία στα αγγλικά και επειδή πάντα έγιναν συζητήσεις στα αγγλικά, νομίζω ότι είναι πιο απλά τα πράγματα. Καταρχάς, θα ήθελα να πω το εξή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εργασία να, σχεδια... να καταρτήσω το σχέδιο αυτό. Γιατί θεωρώ το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το πώς δηλαδή οι μελλοντικοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και κατά δεύτερον, ήταν ενδιαφέρον το θέμα γιατί το ελεγκτικό συνέδριο είχε εκδώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν θα επαναλάβω τα ευρήματα του συνεδρίου, τα βλέπετε άλλωστε και στην έρευνα. Θα τα παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα κατευθείαν να περάσω στις συστάσεις, στα σχόλια τα οποία ε, έχω συμπεριλάβει στο σχέδιο εργασίας μας. Φυσικά καλωσορίζω τη δημοσίευση της έκθεσης, όπως σας είπα, γιατί η απόδοση της ΕΠΣΟ επηρεάζει φυσικά την διαδικασία πρόσληψης, γιατί είναι βασική, το βασικό όργανο για την επιλογή των υποψηφίων. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως, ε, τα θεσμικά όργανα στηρίζονται στην έψο για την ε, κατάρτιση των καταλόγων αυτών για την πρόσληψη. Έχουν και άλλα μέσα, αλλά μέσω της έψο βασικά κινούνται. Και από την έψω εξαρτάται να κάνει αυτή την διαδικασία επιλογής με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό, εξασφαλίζοντας την ισότητα της μεταχείρισης για όλους τους ε, υποψηφίους. Να τονίσω ότι δεν ήταν εύκολο το έργο του συνεδρίου γιατί κατά τη διάρκεια του ελέγχου η ΕΠΣΟ δημοσίευσε και δικό της έλεγχο και μια δική της, ένα δικό της σχέδιο, το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΠΣΟ. Θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο το ελεγκτικό συνέδριο και η έκθεσή του άργησε ε, ένα χρόνο αλλά και ήρθε αν θέλετε ένα χρόνο πολύ νωρίς γιατί δεν ήταν εύκολο αυτό το καθήκον, αυτό, το έργο της έψω. Ε, δεν είχε εφαρμοστεί ακόμα, δεν είχε αξιολογηθεί ακόμα το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα εφαρμοστεί, αλλά φυσικά καλωσορίζω το γεγονός ότι το Ελεκτικό Συνέδριο προσπάθησε να αξιολογήσει το πρόγραμμα αυτό και καλωσορίζω φυσικά και το γεγονός ότι η ΕΠΣΟ προσπάθησε να συμπεριλάβει τις συστάσεις αυτές του Ελεκτικού Συνεδρίου. Φυσικά δεν έχουμε δει ακόμα τον αντίκτυπο του προγράμματος, αλλά είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης η οποία είναι θετική. Φυσικά ορίζω το γεγονός ότι η έψω ε, λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου και γιατί είπα ότι είναι τόσο σημαντικό για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη το πώς επιλέγονται και προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ως εργαλείο επιλογής των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι τελικά θα διαχειριστούν αυτά τα θεσμικά όργανα. Το πώς επιλέγονται οι άνθρωποι αυτοί, το πώς προσλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί, τελικά έχει αντίκτυπο και στην δημόσια εικόνα, στην εικόνα που έχει το κοινό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιλέγονται με αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο τα άτομα αυτά. Και να μην ξεχνάμε ότι τα θεσμικά όργανα αποτελούν και ένα εργοδότη. Με την εικόνα λοιπόν αυτή που προβάλλουν επηρεάζουν και την όλη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στις συστάσεις μου επίσης, καλό να βελτιωθεί η επικοινωνία της έψω με τις δημόσιες αρχές τα κράτη-μέλη για να γίνει ανταλλαγή για τις βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και την ε, διαφήμιση προς το κοινό, δηλαδή τους ενδεχόμενους ε, ενδυνάμει υποψηφίου και για να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες στο, εργατικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον. Γιατί το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα της εργασίας στα ευρωπαϊκά όργανα. Φυσικά καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων γιατί οι εθνικές διοικήσεις ενδεχομένως να έχουν ως στόχο τους ίδιους υποψηφίους όπως και τα όργανα αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί όπως και να έχει αυτός ο συντονισμός σε ό,τι αφορά τώρα την ομάδα των ενδεχόμενων υποψηφίων προς επιλογή Θα ήθελα να κοιτάξουμε και τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια, γιατί θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος των ε, θεσμικών οργάνων μια τέτοια συνεργασία για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση προς τους υποψηφίους και φυσικά με τους αποφύτους προκειμένου και αυτοί να έχουν πιο πολλές πληροφορίες για τις ενδεχόμενες ε, σταδιοδρομίες που θα ακολουθήσουν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο έθιξε και το συνέδριο και το οποίο γνωρίζει εξ ξέρω η ΕΠΣΟ είναι οι γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ των υποψηφίων και μεταξύ των επιτυχόντων. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης. Θα πρέπει να ε, προβούμε στις ανάλογες διαγνώσεις και στις ανάλογες, ε, στα ανάλογα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Λυπάμαι που ούτε στην έκθεση του συνεδρίου, ούτε σε αυτή τη έκθεση στη ΣΕΠΣΟ, δεν αναφέρονται θέματα μεταξύ της μεσαίας και της υψηλότερης διοικητικής τάξης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την γεωγραφική ανισότητα που επικρατεί εδώ. Διαπίστωσα ότι το δείγμα ήταν μάλλον υπερβολικά μικρό για να υπάρχει μια σωστή επισκόπηση. Το δείγμα δηλαδή που ερευνήθηκε. Δεν ε, ήταν δυνατή με τόσο μικρό δείγμα η σωστή αξιολόγηση για την ε, μεσαία και υψηλή διοικητική τάξη. Αλλά νομίζω ότι και εδώ υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες. Πολύ σημαντικό θέμα ήταν ο χρόνος αναμονής. Ο χρόνος δηλαδή που μένουν οι υποψήφοι στην, ε, στους καταλόγους των υποψηφίων. Δηλαδή πολλοί κόσμος περνάει, μπαίνει σε μια λίστα και μετά παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να προσληφθεί. Και αυτό είναι προβληματικό. Και καταρχάς και για τα ίδια τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Αυτό αποτελεί πρόβλημα και για την έψο αλλά και για τα θεσμικά όργανα. Ίσως ε, περιγράφονται με λάθος τρόπο οι ανάγκες. Ίσως οι λίστες ε, να είναι υπερβολικά εκτενείς. Αν είναι τόσο εκτενείς, πολλοί κόσμος ε, τελικά καταλήγει σε άλλες θέσεις εργασίας. Και τελικά δεν υπάρχουν ε, υποψήφοι. Άρα ουσιαστικά χάνεται χρόνος και ενέργεια όταν τελικά αυτός ο κόσμος, αυτά τα άτομα δεν είναι δυνατόν να προσληφθούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να περιμένει ο εργαζόμενος για παράδειγμα χρόνια ολόκληρα. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τους καταλόγους ε, Υπάρχει το θέμα αυτό του χρόνου αναμονή, υπάρχει και το θέμα της διαχείριση των πληροφοριών. Γνωρίζω ότι αυτό το θέμα ξεπερνάει τα όρια του ελέγχου και αν θέλετε ξεπερνάει και τα όρια των δραστηριοτήτων της έψω. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα αυτό της πρόσληψης. Καταρχάς το θέμα τη επιλογής και της πρόσληψης κατά δεύτερο λόγο από τον κατάλογο αυτών των υποψηφίων. Και αυτό νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα θέμα για το κουκουμπού. Να εξεταστεί δηλαδή ο τρόπος πρόσληψης, αν είναι αποτελεσματικός, αν ο τρόπος αυτός πρόσληψης ε, είναι αποδοτικός και αν υπάρχει μια οικονομική, αν θέλετε, ορθότητα. Και επίσης η πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, σε ό,τι αφορά τις διάφορες ε, θέσεις ε, που ανοίγουν. Μου προκάλεσε τέτοια έκπληξη το γεγονός ότι οι υποψήφοι οι οποίοι τελικά έχουν περάσει και έχουν μπει σε μια λίστα δεν ενημερώνονται για τις ε, θέσεις αυτές εργασίας που ανοίγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί στην τελική ανάλυση το θέμα είναι να γίνεται μια καλή επιλογή και μια σωστή πρόσληψη των σωστών ατόμων. αναρωτιέμαι κατά πόσο θα λύσει το πρόβλημα η απόσπαση εργαζομένων από άλλους, υπαλλήλων από άλλους ε, τομείς, από άλλα φυσικά όργανα στην ΕΠΣΟ. Δεν έχει εφαρμοστεί με το σύστημα αυτό, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα επιδράσει, αλλά θεωρώ ότι ίσως να είναι υπερβολικό το διάστημα των τεσσάρων ετών απόσπασης για να γίνει αν θέλετε πιο έντονος ο σύνδεσμος, η σύνδεση μεταξύ της έψο και του ε, οργάνου από το οποίο προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί αποτελεί πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο. Κάποιες πιο τεχνικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά δηλαδή ενδεχόμενε ασάφειε στι προκηρύξει των διαγωνισμών. Αυτέ θα πρέπει να αποφεύγονται. Γι' αυτό λοιπόν Καλό την έψω να καταστήσει πιο απλές ε, αυτές τις προκηρύξεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται επανελειμμένες ε, διορθώσεις των προκηρύξεων, να μην ξέρουν οι υποψήφοι τελικά ποια κριτήρια ισχύουν. Επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα μετάφρασης. Ε, ξέρω ότι μάλλον πολλά από τα προβλήματα προέρχονται από τη μετάφραση. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τις προκηρύξεις αυτές. Επίσης, σημαντικό είναι να βελτιωθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Να είναι σαφές δηλαδή πώς μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις οι υποψήφοι γιατί σε διάφορες διοικητικές, σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες ε, ε, ο υποψήφιος ε, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει η να το εξετάσει για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν διάφορα σώματα σε ό,τι αφορά την υποβολή ενστάσεων. Δεν ξέρω αν είναι κοινή πρακτική αυτό ή αν ήταν κάτι το εξαιρετικό, αλλά συνέβη το εξής. σε διάφορες διαδικασίες ενστάσεων να είναι το ίδιο άτομο αυτό το οποίο εξετάζει τις διάφορες φάσεις μιας ένστασης. Αυτό φυσικά δεν είναι δυνατόν. Επίσης στο μέλλον θα ήθελα να διδαχτούμε από διάφορες ε, υποθέσεις ε, δημόσιων υπαλλήλων κατά της ΕΠΣΟ. Και όπως αναφέρει το λεκτικό συνέδριο, στο σημείο αυτό η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η υπερβολικά μακροσκελής διαδικασία επιλογής. Θα σταματήσω εδώ. Όπως σας είπα, ελπίζω αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για την, ε, της περαιτέρω συζήτησής μας. Ξέρω ότι η έκθεση εστιάζεται σε θέματα επιλογής, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσουν τα θέματα επιλογής και πρόσληψης. Και να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ελπίζω και η Κοκομπού κάποια μέρα θα εξετάσει τα θέματα πρόσληψης, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ε, των δημοσίων υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την πολύ καλή και πολύ εκτενή έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαιρετικούς υπαλλήλους σε όλους τους τομείς, αλλά η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι να έχουμε τους βέλτιστους. Με τον τρόπο που τώρα προσλαμβάνουμε δεν το επιτυγχάνουμε. Είναι δύσκολη διοργάνωση, ξεκινάμε την επιλογή, ε, δεν υπάρχει μία ενιαία επιλογή είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ δαπανηρή και όπως ξέρουμε και σε πολλά πανεπιστήμια ε, ε, πολλές ε, φορές απλώς ξεκαθαρίζει κανείς αλλά έτσι δεν έχουμε τους καλύτερους διότι είμαστε ένας πολιτικός οργανισμός που χρειάζεται πολιτική κατανόηση διότι χρειάστηκε μία φορά να ε, αναλύσω μία ομιλία που την οποία ε, ε, εγώ είχα γράψει ήμουνα τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν κατάλαβα τη λογική μου δηλαδή με την καλύτερη θέληση δεν τα κατάφερα αυτό σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνουμε την επιλογή των καλυτέρων και πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε τις μεθοδολογίες μας επίσης υπάρχουν μήνες και χρόνια που παραμένουν οι επιτυχώντες τους καταλόγους και χάνετε τους καλύτερους. Και εδώ δεν αναφέρουμε μόνο στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο αλλά και στην ε, πολύ ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Τράπεζα η οποία επίσης προσλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η τράπεζα έχει διαφορετική ε, διαδικασία η οποία εστιάζεται πολύ περισσότερο στο τραπεζικό τραπεζικό σύστημα και μπορούμε να διδαχθούμε πολλά. Και ε, δεν ε, φεύγουν πολλοί διότι παραμένουν στη λίστα πάρα πολύ χρόνο ακόμη και αν πρόκειται να πληρωθούν πολύ καλά. Ξέρουμε δηλαδή ότι οι υποψήφοι οι οποίοι απευθύνονται εις ε, τους ε, γενικούς διευθυντές για να επιλεγούν βάσει ε, του καταλόγου έχουν καλύτερες ε, πιθανότητες να προσληφθούν γρήγορα. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το, στην, το, Ευρωπαϊκό, το Ελεκτικό Συνέδριο στην τρίτη του επιλογή αναφέρθηκε στο γλωσσικό. Και εδώ θα ήθελα να μου πει ο εκπρόσωπος της ΕΠΣΟ είναι το ε, διαψεύσει ότι τα γερμανικά που είναι η τρίτη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η τρίτη γλώσσα δηλαδή υπάρχει διάκριση εναντίον των γερμανικών πρώτα είναι ε, τα, τα αγγλικά μετά τα γαλλικά μετά τα γερμανικά κάποιος που ξέρει ε, γαλλικά και γερμανικά μόνο και όχι αγγλικά δεν έχει καμία δυνατότητα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις περιπτώσεις και τις γνωρίζω τότε πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια. Πρέπει να πούμε τη μητρική, τα αγγλικά και μία δεξιότητα όπως το λέει το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή τη δυνατότητα να μάθει κανείς μία άλλη γλώσσα γρήγορα. Αν τώρα όμως ε, είμαστε σε ισότιμη αξιολόγηση των τριών γλωσσών πρέπει να σας πω ότι η έψο τουλάχιστον ε, για τα γερμανικά δεν συμπεριφέρεται δίκαια και πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια αυτά γιατί νομίζω ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα επικοινωνίας ας ξεχάσουμε ε, τους τσακωμούς τα αγγλικά είναι η γλώσσα επικοινωνίας πρέπει όμως να αναγράφεται διότι υπάρχουν εξαιρετικοί ε, υποψήφοι οι οποίοι μπορούν να εκφραστούν σε μια άλλη γλώσσα αλλά όχι αγγλικά και τότε δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν έχουμε σωστά κριτήρια. Ε, μόνο έτσι θα μπορούμε να βρούμε τους καλύτερους τους οποίους χρειαζόμαστε. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε τα κριτήρια και να τα αναθεωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότησή του. Την εισηγήτρια μάλλον. Θα ήθελα να τονίσω μερικά προβλήματα που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Το ελεγκτικό συνέδριο κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Συγκρίνει την, ε, ε, κάνει μάλλον τον απολογισμό της αποτελεσματικότητας σε βάση των κριτηρίων. Αλλά αυτά τα κριτήρια είναι καλά. Λέγεται στην έκθεση ότι ο τριετής σχεδιασμός είναι ένα κριτήριο το οποίο δεν εφαρμόζεται πάντα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε το χρόνο, πρέπει να μειώσουμε την διαδικασία μέχρι 9 μήνες. Οπότε αν τα λέμε όλα αυτά, ο σχεδιασμός πάνω στα τρία χρόνια είναι απαραίτητος, διότι τότε η διαδικασία δεν θα είναι καν ε, χάνει όλη τη τη δυναμική. Τώρα, για τους επιτυχόντες. Ορισμένα κριτήρια είναι σαφή. Ένα τρίτο των υποψηφίων πρέπει να πετύχουν αλλά αν εμείς εξετάσουμε και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, βλέπουμε ότι δεν προσλαμβάνεται πάνω από το 10% που έχουμε στους καταλόγους. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε εμείς μια μεγαλύτερη συμμετοχή στους διαγωνισμούς έψω, χρειάζεται και μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ξέρουμε ότι έχουμε προβλήματα, ας πούμε για τους διερμηνείς των νέων κρατών μελών. Αντί λοιπόν εμείς να ξοδεύουμε λεφτά και μέσα, θα πρέπει αυτά τα κονδύλια να τα αφιερώσουμε στην κατάρτιση ατόμων που μετά μπορούν να διοριστούν. και πρέπει να δούμε μετά πώς γίνεται και η γεωγραφική κατανομή μέσα στην αναλογία δηλαδή των επιτυχόντων και των προσληφθέντων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη φίγουρα και η γεωγραφική κατανομή. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. και των κρατών μελών και των πολιτών τους. Αυτός ο συσχετικοσμός δυνάμεων πρέπει να αλλάξει, διότι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια της γεωγραφικής αντιστοιχίας να λάβουμε υπόψη μας και άλλα κριτήρια. Τώρα για τις διαδικασίες πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια διότι θέλουμε πολύ εξειδικευμένους και ικανούς επαγγελματίες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περιμένουν ένα χρόνο ή δύο χρόνια μέχρι να τους δοθεί μια απάντηση για, να, για το αν θα διοριστούν ή όχι. Η διαδικασία για παράδειγμα να μην κρατάει πάνω από 9 μήνες και αυτή η διαδικασία να είναι διαφανής να μπορούν οι υποψήφοι να ενημερώνονται σε όλες τις φάσεις της επιλογής. Και τελευταίο οι δαπάνες και το κόστος της πρόσληψης. Εμείς έχουμε 7.100 ευρώ αυτό είναι το κόστος ενός επιλεγμένου υποψηφίου. Η έψο συστήνει να αυξήσουμε αυτό το κόστος για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση και δημοσιοποίηση. Πρέπει να ελέγξουμε όμως εμείς τις δαπάνες και το κόστος για να έχουμε ένα πραγματικό συσχετισμό ε, ποιότητας και απόδοσης. Ευχαριστώ. Έχω, μία, έχω ερωτήσεις για τον επικεφαλής της ΕΠΣΟ που είναι εδώ. Είναι περίεργο πως οι στατιστικές μας λέγουν ότι ορισμένες χώρες είναι πιο επιτυχείς από άλλες. Ξέρουμε βέβαια πόσο, πώς παρακολουθούν οι χώρες ε, ε, αυτά τι στατιστικές. Οι Βέλγοι έχουν 22% ε, έχουν περισσότερους υποψηφίους από ότι η Ιταλία ή η Γερμανία οπότε γιατί οι Βέλγοι είναι πιο επιτυχής από όλους τους υπολείπους. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Μετά, η αντικειμενικότητα ή μάλλον η διαδικασία η οποία προτείνεται εδώ για την επιλογή των υποψηφίων είναι πολύ αντικειμενική ή τουλάχιστον τονίζεται η αντικειμενικότητα. Μετά όμως καταρτίζεται ένας κατάλογος πιθανών υποψηφίων για πρόσληψη και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι πώς οι υπηρεσίες, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι υπόλοιποι, πώς επιλέγουν από τον κατάλογο αυτό. Θα ήθελα να έχω μία αξιολόγηση για το πόσο αντικειμενική είναι αυτή η διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι ε, κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται. Ε, και αυτό ίσως απαντά στο θέμα των ε, Βέλγων υποψηφίων και τις επιτυχίες τους. Ε, δηλαδή πώς καταλήγει κανείς από τον κατάλογο να βρεθεί σε μια πραγματική θέση εργασίας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον υπεύθυνο της ΕΠΣΟ που είναι παρόν. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση του. Καλώς ορίζω την έκθεση αυτή. Δεν ήταν εύκολη η χρονική συγκυρία, αλλά παρόλα αυτά αποτέλεσε χρήσιμη συμβολή για την έψο. Είναι μάλλον ε, ασυνήθιστη η κατάσταση, γιατί καλωσορίζουμε και δεχόμαστε φυσικά τις συστάσεις του συνεδρίου, αλλά έχουμε ήδη εφαρμόσει αρκετές εξ αυτών και όσες δεν τις έχουμε εφαρμόσει θα τις εφαρμόσουμε στο εγγύης μέλλον. Έχουμε εφαρμόσει ένα ε, εκτενές πρόγραμμα προσαρμογής στην ΕΠΣΟ, το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο. Πολλοί βουλευτές κάναν διάφορα σχόλια με τα οποία συμφωνούμε. Μιλάμε για το μέλλον της ποιότητας των ευρωπαϊκών ε, υπηρεσιών. Θεωρώ ότι ένα πρόγραμμα το οποίο, ένα σχέδιο το οποίο είναι 50 χρόνια ε, παλιό, αν θέλετε, είναι και κατά 50 χρόνια παροχημένο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι όχι να αυξήσουμε το κόστος, να αυξήσουμε όμως την αποτελεσματικότητα γιατί θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσελκύουμε τους καλύτερους και να επιλέγουμε τους καλύτερους εξ αυτών. Και αυτό που είναι σημαντικό για το μέλλον, ακόμα και αν ε, μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε την πρόκληση της διεύρυνσης είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Θα υπάρξει σε όλα τα όργανα μια αλλαγή γενιάς, αν θέλετε, σε όλα τα θεσμικά όργανα. Γιατί πολλοί θα φύγουν στη σύνταξη τα επόμενα δέκα χρόνια και αυτό αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα έντονο στο Κοινοβούλιο και παράλληλα τα δημογραφικά στοιχεία σε όλη την Ένωση καταδεικνύουν, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί ταλαντούχοι απόφοιτοι τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπιστούν ε, οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία επιλογής η οποία δεν θα είναι μόνο γρήγορη και αποτελεσματική αλλά και σύγχρονη. Δεν, ε, μπορούμε να έχουμε παροχημένες τέτοιες μεθόδους γιατί με τις μεθόδους αυτές δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας επαρκώς στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τα καλύτερα ταλέντα. Γι' αυτό λοιπόν αναζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλούς ε, τέτοιους ε, θεσμικούς οργανισμούς στα κράτη-μέλη, αλλά και σε διεθνείς οργανώσεις Μάθαμε από τις εμπειρίες αυτές και θεωρώ ότι τα μέτρα που προτείναμε και τα οποία εφαρμόζουμε εν μέρη ήδη θα μας καταστήσουν ικανούς για να προσελκύσουμε όντως τους καλύτερους και να επιλέξουμε τους καλύτερους, να κοιτάξουμε κάποια θέματα. Να κάνω κάποια σχόλια. σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Όντως θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να περάσουμε πέρα από τη φούσκα των Βρυξελών και του Λουξεμβούργου. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει άμεση σύγκρουση συμφερόντων, θα έλεγα, με τα κράτη-μέλη, γιατί και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να διασφαλιστεί ότι ένα τμήμα των πλέον ταλαντούχων ε, εργαζομένων τους θα καταλήξουν στα θεσμικά όργανα και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Άρα συνεργαζόμαστε με αρκετά κράτη-μέλη για να διασφαλιστεί και έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη και ελπίζουμε όντως να περνάει το μήνυμα αυτό. Εφαρμόζουμε στρατηγικές βάσει χωρών και συγκεκριμένων αναγκών και επίσης ε, απευθυνόμαστε και προς τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Συμμετέχουμε σε διάφορες ε, οργανώσεις πανεπιστημιακών ε, κύκλων στο Λονδίνο, στη Γερμανία. Συνεργαζόμαστε λοιπόν ε, τα πανεπιστήμια. Και επίσης το γεγονός ότι έχουμε πλέον την ιστοσελίδα μας σε 23 γλώσσες και ότι οι προκηρύξεις γίνονται σε 23 γλώσσες πλέον, αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα βελτίωση. Και πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση. Το θέμα της γεωγραφικής ανισότητας που παρατηρείται, νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις στο σημείο αυτό. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια ήταν η κλασική περίπτωση λόγω της διεύρυνσης. Γιατί εστιαστήκαμε ασφαλώς, εντονότατα, στα θέματα των νέων κρατών μέλων. Αυτό θα αλλάξει τα επόμενα 5 χρόνια. Και επίσης ε, έγιναν και κάποια σχόλια για το πόσο ε, είναι ελκυστική η μισθή στα διάφορα θεσμικά όργανα και αυτό φυσικά εξαρτάται από το κράτος μέλος το οποίο εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος γιατί σε κάποια κρατημέλη είναι δύσκολο να προσελκυστούν οι υποψήφοι σε άλλα, σε άλλα κρατημέλη υπάρχουν θέματα ανεργίας και όλα αυτά φυσικά είναι σημαντικοί παράγοντες για το πόσο ελκυστικές οι θέσεις εργασία μας και φυσικά χρειάζεται πιο πολύ δουλειά στους ε, στα κράτη-μέλη εκείνα όπου είναι όλοι οι παράγοντες αρνητικοί. Υπάρχει συνδυασμός δηλαδή αρνητικών παραγόντων. Για την επιλογή τώρα των αποφύτων έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Αλλά αυτό ίσως να υπερβαίνει κάπως, αν θέλετε, και τις δικές μου αρμοδιότητες στην έψο, γιατί άπτεται πιο πολύ θεμάτων πρόσληψης. Τώρα, αν οι συγγνώμη, οι επιλεγμένοι, αυτοί που έχουν μπει στη λίστα, οι επιτυχώντες, ε, ενημερώνονται σωστά. Αυτά λοιπόν αποτελούν προβλήματα σημαντικά. Και φυσικά τίθεται και το θέμα και του χρόνου αναμονή των επιτυχόντων στι λίστε. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό ανάπτυξη, το ADP, θα, θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό προκειμένου ο αριθμός των επιτυχόντων να είναι πιο κοντά στον αριθμό των προσλήψεων τα επόμενα χρόνια. Και αυτό γίνεται πιο σαφές και από τις δημοσιονομικές προοπτικές και έτσι στο μέλλον θα διασφαλιστεί ότι το να είναι κανείς ε, επιτυχών συνεπάγεται ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να προσληφθεί. Καταλαβαίνω τις αμφιβολίες που επικρατούν για την απόσπαση των ε, υπαλλήλων στην έψο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό και αποτελεί και το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Γιατί το να υποχρεώσουμε κάποιους υπαλλήλους να φύγουν κάποιες ημέρες ή κάποια, ε, κάποιες εβδομάδες ε, από τη δουλειά τους δεν θεωρώ ότι θα λειτουργήσει η απουσία μελών ε, των επιτροπών αυτών αποτελεί ένα βασικό λόγο καθυστέρησης. Κατά δεύτερον, δεν θα υπάρχει συνέχεια. Κάθε Συμβούλιο Επιλογής θέτει δικά του κριτήρια, αλλάζει τη σύνδεση κάθε φορά. Οι υποψήφοι δεν ξέρουν πού τύφεται ο πύχης. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη συνοχής δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ε, θεσμικών οργάνων, που είναι επίσης πολύ διαφορετικές. Και επίσης δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να αφήνονται τα θέματα αυτά επιλογής στα χέρια ερασιτέχνων ουσιαστικά, όσο ταραντούχη κι αν είναι αυτή. Άρα θεωρώ ότι ο τρόπος αυτός με την απόσπαση αποτελεί ε, τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης αδυναμίας. Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη διαγωνισμών έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, ριζικές αλλαγές όχι μόνο το γεγονός ότι διατίθενται σε 23 γλώσσες, αλλά πλέον υπάρχει και ένας τυποποιημένος οδηγός, ο οποίος ε, μεταφράζεται μία φορά, είναι πολύ σαφής και τροποποιείται στην παρούσα φάση για να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι δέχουσες αλλαγές. Θα είναι πολύ πιο συνοπτικός και θα παρουσιάσει με καλύτερο τρόπο τις διαδικασίες ε, προκήρυξη διαγωνισμός και ελπίζουμε αυτό να μειώσει τα λάθη. Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε τέσσερις ε, μηχανισμούς ε, υποβολής ένστασης και τα διευκρινίζουμε αυτά σε κάθε υποψηφίο. Και κάνουμε έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να μην είναι τα ίδια τα άτομα εκείνα τα οποία εξετάζουν και αξιολογούν ένα αίτημα για επαναξιολόγηση μιας υποψηφιότητας με τα άτομα εκείνα τα οποία τελικά αποφασίζουν. Και γενικώ παρατηρήθηκε 40% μείωση των ενστάσεων προς την έψο και 60% μείωση αναφορικά με υποθέσεις ε, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά εκπληκτική αυτή η εξέλιξη και αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι ε, έχουμε εφαρμόσει αυτά τα μέτρα για να αντιμετωπίζουμε με καλύτερο τρόπο τους πελάτες μας όπως θεωρούμε και να αντιμετωπίζουμε με καλύτερο τρόπο ε, τα προβλήματά τους. Να μιλήσω τώρα γερμανικά σε ό,τι αφορά την κριτική για τα γερμανικά και την διάκριση που υπόκεινται. Θα ήθελα να σας πω ε, ότι σε ό,τι αφορά την έψοδο δεν υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Έχουμε πλέον τρι... μάλλον, ε, διαδικασία επιλογής σε τρεις γλώσσες όπου εξισώνονται τα αγγλικά, γαλλικά και τα γερμανικά. Δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση κατά της γερμανικής γλώσσας. Όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει να κάνουν την διαδικασία επιλογής στη δεύτερη γλώσσα τους, τα αγγλικά τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Συμφωνώ με το στόχο, με το ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε τους καλύτερους ε, από όλη την Ευρώπη, γιατί αν ε, δεν τους προσελκύσουμε θα έχουμε προβλήματα όλοι μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε μόνο τεστ ε, λογικής γνώσεων, αλλά να ελέγχουμε και τις ικανότητες των υποψηφίων. Και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, το μύτο που διατρέχει όλο το πρόγραμμα ανάπτυξης αυτό της ε, ΕΠΣΟ. Θέλουμε και τεστ λογικής, όχι μόνο λογικής όμως. Αν έχουμε δηλαδή 10, 20, 30 χιλιάδες υποψηφίους, θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε μια προκαταρτική επιλογή Νομίζω ότι στα αγγλικά το λέμε αυτό self-assessment, δηλαδή να δουν και οι υποψήφοι τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, τι συμπεριλαμβάνει κάθε θέση εργασίας για να μπορεί να κάνει και κάθε υποψήφιος μια δική του πρώτη αξιολόγηση. Αυτό θα ενισχυθεί ως διαδικασία από το 2010, αυτό δηλαδή το στοιχείο της αυτοεπιλογής, της αυτοαξιολόγησης. Και επιμένω ότι ε, ελέγχουμε και αξιολογούμε τις εικονότητες σε ό,τι αφορά την γεωγραφική ισότητα. Γιατί σημειώνουν τέτοια επιτυχία οι Βέλγοι στις διαδικασίες επιλογής μας. Καλή ερώτηση. Ίσως θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και άλλους συναδέλφους. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ένα μέρος της όλης ε, λύσης είναι ότι είναι τόσο εξειδικευμένες οι διαδικασίες επιλογής, τα τεστ γνώσεων και το καθεξής που Τι να σας πω, υπάρχουν μαθήματα από τα συνδικάτα των ε, ε, θεσμικών οργάνων, αλλά και από την ελεύθερη αγορά. Εκατοντάδες βιβλία για το πώς περνάει κανείς τις διαδικασίες επιλογής της έψος και τα μαθήματα αυτά, τα βιβλία αυτά ουσιαστικά διατίθενται στον κόσμο που μένει στο Λουξεμβούργο ή στο, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Και εδώ υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση. Και αυτό θα επιληθεί στο μέλλον, γιατί δεν θα ελέγχονται οι γνώσεις, δεν θα υπάρχουν πλέον 250 ερωτήσεις. Όχι. Θα ελέγχουμε τις ικανότητες των ε, υποψηφίων. Και αυτό νομίζω ότι θα αποτελέσει μια πολύ σωστότερη βάση επιλογής. Σωστό είναι ότι και ε, οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις θέσεις, αλλά και αυτό υπερβαίνει τις αρμοδιότητές μου. Ξέρω ότι έχει προτείνει τέτοια μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δυστυχώς δεν συμφωνούν όλα τα θεσμικά όργανα. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να το, θυμί... το συζητήσει το θέμα αυτό το... η Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο μας ε, στις 18 Σεπτεμβρίου. Και τώρα να περάσω και πάλι στα αγγλικά για τις υπόλοιπες ερωτήσεις που τέθηκα για την ε, τριετή περίοδο προγραμματισμού. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητη και νομίζω ότι και με τις αντατήσια προγράμματα θα αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα στη διαδικασία επιλογής και στις κατεπήγουσες ανάγκες πρόσληψης σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ατόμων που προσλαμβάνονται νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από το 10% για τους ε, επαγγελματίες με τα σωστά προσόντα φυσικά θα είναι και πιο σύντομος ο χρόνος αναμονής και θέλουμε να διοργανώνουμε και να ολοκληρώνουμε διαγωνισμούς μεταξύ 5 και 9 μηνών. Για τους εξειδικευμένους επαγγελματίες θα είναι ακόμα μικρότερος ο χρόνος αυτός. Επίσης θα θέλουμε να βελτιώσουμε τις προκηρύξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εξειδικευμένες θέσεις όπως αυτές των διερμηνέων. Δεν ήταν πάντα εύκολη αυτή η ενημέρωση για τις προκηρύξεις και νομίζω ότι αν ε, δεν συντονιστούμε, αν δεν συνεργαστούμε και αν ε, ε, παραμείνει αυτό σε επίπεδο θεσμικού οργάνου, δεν θα υπάρξει αντίκτυπο σημαντικό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να έχει αντίκτυπο η δράση μα στη διεθνή αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα την αύξηση του κόστου, ξέρουμε ποιο είναι ο προπολογισμό μα και θα προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε αυτόν. γιατί κατά τα άλλα δεν θέλουμε να αυξηθεί το κόστος της διαδικασίας επιλογής. Ανά ε, το κόστος των 7.000 ευρώ που ισχύει κατά μέσο, όρος, κατά μέσο όρο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. για να μην συζητήσω το κόστος του να προσλάβουμε το λάθος άτομο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να απολυθεί. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή επένδυση για να γίνει σωστή πρόσληψη εξ αρχής και νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο προκειμένου να είναι η διαδικασία επιλογής πιο αποτελεσματική και πιο σωστή και πιο οικονομική στο μέλλον. Δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση 11 κάθετος 2009. Ε, αηφορία και υποστήριξη των σχέδιων Life, των σχεδίων Nature εκ μέρου επιτροπή. Επιτροπής. Το λόγο έχει ο κύριος Καζαμίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη μας επαφή από τον καιρό της ε, εκλογής σας ε, τον τελευταίο καλοκαίρι ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ όπως και στην εισηγήτρια του θέματος και σε όλους τους νέους βουλευτές κάθε επιτυχία στο έργο σας. Και σε όλους τους επανεκλεγέντες επίσης βουλευτές καλή δύναμη έτσι που όλοι μαζί να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας για το καλό της κοινότητας και των λαών των κρατών μελών μας. Ε, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι αρκετοί βουλευτές ε, είναι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω ετοιμάσει και τη σημερινή παρουσίαση για το θέμα που μας απασχολεί ανάλογα. Το live λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον. Η διαχείριση του ασκείται απευθείας από την Επιτροπή και από οικονομική άποψη πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που είναι ειδικά αφιερωμένο στο περιβάλλον. Συνεπώς, αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρώτα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από το LIFE ξεκίνησαν το 1992 και οι χρηματοδοτήσεις LIFE για σχέδια συνεχίστηκαν στο πλαίσιο των μεταγενέστερων ειδικών μέσων LIFE έως την τρίτη φάση, που είναι γνωστή ως LIFE 3, για την περίοδο 2000-2006. Η χορήγηση για το LIFE 3 ανήλθε σε 957 εκατομμύρια ευρώ και με τη νέα φάση του LIFE, που ονομάζεται LIFE SIN διατίθενται 2 δισεκατομμύρια 143 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2013. Στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης που άσκησε η Επιτροπή όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν για τα σχέδια του LIFE 3, δηλαδή για την περίοδο 2000 μέχρι το 2006. Φύση, κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου των σχεδίων, από την άποψη της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των σχεδίων. Επίσης, διενεργήθηκε ταυτόχρονα έλεγχος σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για το νέο Life Sin, δηλαδή για την περίοδο που επακολουθεί ξεκινώντας από το 2007 μέχρι το 2013. Και οι παρατηρήσεις του συνεδρίου παραμένουν σημαντικές για τη νέα περίοδο, δεδομένου ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας που θίγονται αφορούν και το νέο σχέδιο Life Sin. Κατά την περίοδο λοιπόν 2000-2006 χρηματοδοτήθηκαν από το Life ε, Φύση 434 σχέδια τα οποία υλοποιήθηκαν σε 26 κράτη-μέλη με συνολικό ποσό 436 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου ε, επιδοτήθηκαν με κοινοτικά κονδύλια 1 εκατομμύριο ευρώ ανά κάθε σχέδιο στο σκέλος φύση και βιοπικιλότητα διατίθεται ποσό 850 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013, δηλαδή περίπου διπλασιάζεται το ποσό. Πράγματι, το Life Φύση συγχρηματοδοτεί σχέδια στα κράτη-μέλη, κυρίως σε σχέση με το δίχτυ Natura 2000, με σκοπό τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων. Τα σχέδια αυτά πρέπει να προσδίδουν προς τη θέμενη αξία όσον αφορά την επίδειξη και να συμβάλλουν στη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής ως προς τις μεθόδους και τους τρόπους προσέγγισης σχετικά με τη διατήρηση. Οι προκατακτικές ελεκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν σύντομα ότι η εποπτεία και διαχείριση του life φύση αποτελούν όχι εύκολη αλλά πολύπλοκη διαδικασία δεδομένου ότι τα χρηματοδοτούμενα σχέδια επηρεάζονται από διαφορετικές καταστάσεις στους διάφορους τόπους σε ολόκληρη την Ένωση, υλοποιούνται από διάφορα είδη δικαιούχων, πρέπει να έχουν διαρκή αντίκτυπο στη διατήρηση διαφόρων ειδών και οικοτόπων και τέλος πρέπει να προσδίδουν απαραίτητα προστιθέμενη αξία μέσω της διάδοσης των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων, δηλαδή τα διδάγματα που αντλούνται και βέλτιστες πρακτικές που επισημαίνονται. Από το 1992 που ξεκίνησε το πρόγραμμα και εξή, η η Επιτροπή ανέπτυξε και βελτίωσε σταδιακά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προγενέστερων ελέγχων του συνεδρίου και ιδιαίτερα της ειδική έκθεσης αριθμός 11 από το 2003. Τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου συγκεντρώθηκαν από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και μέσω επισκέψεων για την εξέταση 35 σχεδίων σε 6 κράτη-μέλη, το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εξωτερικές ομάδες παρακολούθησης και επικοινωνίας, στους αξιολογητές των σχεδίων και στο θεματικό κέντρο για τη βιολογική ποικιλότητα που ενεργεί στα πλαίσια σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος δεδομένου ότι έχουν στενή εταιρική σχέση με την Επιτροπή για τη Διαχείριση και την Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Θεμάτων. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές τα σχέδια που ελέγχθηκαν συνέβαλαν στη διατήρηση των στοχοθετημένων ειδών και οικοτόπων, ιδίω του τόπου Natura 2000, ενισχύοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών και στηρίζοντας τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την εθελοντική εργασία και τη δέσμευση των ενώσεών τους υπέρ της διατήρησης της βιοπικιλότητας. Ωστόσο, επισημάνθηκαν οι ακόλουθες ανεπάρκειες σε σχέση με τις διάφορες φάσεις της διαχείρισης των σχεδίων, οι οποίες επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους. Στη διαδικασία επιλογής δόθηκε ασαφής και μειωμένη βαρύτητα στους σχετικούς παράγοντες βιωσιμότητας, κατά τη βαθμολόγηση των, σχεδίων, των σχεδίων για το Life Plus και η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επιχορηγήσεις τα χρονοβόρα. Στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή την υλοποίηση και την παρακολούθηση, δεν αφιερώθηκε επαρκής προσοχή στα αποτελέσματα των σχεδίων και οι συμβάσεις και τα σχέδια διαχείρισης ούτε εγκρίνονταν ούτε εφαρμόζονταν συστηματικά στη διάδοση των αποτελεσμάτων, στην τρίτη φάση της όλης διαδικασίας, δεν τίθοντο συστηματικά στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού εκτός του άμεσου περιβάλλοντος του σχεδίου, είτε αυτό ήταν η περιφέρεια σε μια χώρα ή σε μια ολόκληρη χώρα, συναφείς πληροφορίες με δυνητική προστιθέμενη αξία σχετικά με επιμέρους σχέδια όσον αφορά τα διδάγματα που αντλούνται, τις βέλτιστες πρακτικές που επισημαίνονται, και τις λεπτομέρειες τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες που αποκτώνται. Και τέλος, στην τέταρτη και τελευταία φάση της όλης διαδικασίας, στη μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δηλαδή, η Επιτροπή διαθέτει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων σχεδίων, δεδομένου ότι δεν έχει καθιερωθεί καμιά εκ των υστέρων διαδικασία παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων σχεδίων και δεν έχει καθιερωθεί σειρά ενδεδειγμένων δικτών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυχάνονται. Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από τη θέσπιση του ΛΑΙΦ το 1992, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Επιτροπής, προκειμένου να αποκομίζεται η βεβαιότητα ότι τα μέτρα διατήρησης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυχάνουν καλύτερα τους στόχους τους και συνεχίζουν να είναι βιώσιμα όταν σταματήσει η κοινοτική χρηματοδότηση του σχεδίου. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι εγκρίνονται και εκτελούνται μόνο οι κατάλληλα εκπονηθήσεις προτάσεις σχεδίων. Επίσης, πρέπει να επιμένει στην καθιέρωση κατάλληλων οργανωτικών και χρηματοοικονομικών δομών, ώστε τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδια να έχουν διαρκή αντίκτυπο. Συνιστάται λοιπόν στην Επιτροπή να δώσει περισσότερη βαρύτητα στους διάφορους παράγοντες που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των σχεδίων, να βελτιώσει τη διάδοση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και να καθιερώσει συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων μετά την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κλείσω τη σύντομη παρέμβαση μου εκφράζοντας τις ευχαριστίες τόσων εμού όσων και των συνεργατών μου για την πρόσκληση εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στην εισηγήτρια για την εξαίρετη συνεργασία μαζί της και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και τον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος αποδέχτηκε πολύ επικοδομητικά τα ευρήματα του ελέγχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάννα Ιβάνοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ αγγλικά, διότι ε, έλαβα την ε, τελευταία στιγμή ε, τα έγγραφα, δεν μπόρεσα να μεταφραστούν και όλη μου η δουλειά έχει γίνει αγγλικά. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ σαφή έκθεσή του και τις συστάσεις. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό και Επίσης ο χρόνος ήταν περιορισμένος διότι όπως ε, λέχθη τα, κοιτάξαμε ε, προγράμματα ε, πολλών εκατομμυρίων ευρώ δηλαδή 957 εκατομμυρίων ευρώ για το LIFE 3 και το νέο πρόγραμμα ήταν 2 δισεκατομμύρια 143 εκατομμύρια ευρώ για το 2007-2013. Ε, ήταν ε, λοιπόν πολύ σημαντικό και προτού καταλήξω εις τις ε, συστάσεις ε, και στα συμπεράσματα θέλω να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη έκθεση η οποία γίνεται. Μία τέτοια έκθεση είχε ήδη καταρτιστεί το 2003 για να ε, εντοπίσουμε τις αδυναμίες στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μορφώθηκε με πολλές από τις συστάσεις τα επόμενα έτη αλλά ε, το 2004 στην έκθεση λέγεται ότι όλες οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είχαν ληφθεί υπόψη για να μπορέσει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πόρων εξετάσαμε τέσσερις φάσεις. Πρώτον τη διαδικασία επιλογής, δεύτερον την εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος, τρία η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και τέσσερα μακροχρόνια διαχείριση των συμβολέων. Τα θέματα αυτά έχουν επαναληφθεί πολλές φορές και ουσιαστικά είναι η πεμπτουσία του ελέγχου και της εκθέσεως αυτής. Γι' αυτό και θέλω να διευκρινίσω ότι πρέπει να καθορίσουμε την αηφορία διότι βασίζεται σε οδηγίες βάσει των οποίων καταρτίστηκε και η έκθεση. Ένα βασικό στοιχείο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν το πρόγραμμα μπορεί να αποκαταστήσει την ε, ε, διατήρηση και την κατάσταση και την διατήρηση των ειδών. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Δεύτερο είναι το θέμα χρόνου πρόκειται να συνεχίσει το πρόγραμμα ε, πιο μακροπρόθεσμα και να μπορέσει να διχειριστεί εγκαταλελειμμένα ήδη. και τέλος υπάρχουν διάφορες λειτουργίες για την μακροχρόνια διαχείριση του προγράμματος που είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση του προγράμματος διότι αν κοιτάξουμε παραδείγματος χάνει τη διαδικασία επιλογής θα διαπιστώσουμε ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αποδίδει μεγάλη σημασία στα προγράμματα Life Sin και μία μακριά διαδικασία μέχρι ότου μπορέσει να ληφθεί απόφαση. Ε, δεν ε, μπόρεσαν να ε, εφαρμοστεί επαρκώς η απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων δεν υπάρχει συστηματική αποδοχή των προγραμμάτων της διοίκησης όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Λοιπόν, δεν ήταν επαρκής και ε, για την μακροχρόνια διαχείριση ε, έπρεπε ε, να μπορέσει κανείς να εγκαταστήσει μία υπόγεια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού για να αξιολογήσει την αποδοτικότητα της υπέργειας η οποία όμως πλέον δεν χρησιμοποιείται. Οπότε η σύσταση θα έπρεπε ε, να ήταν ότι δεν έπρεπε να έχει χρηματοδοτηθεί η αντικατάσταση των αχρήστων γραμμών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που αναφέρω για να σας πω ότι η διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά. Μετά, όσον αφορά την ε, ε, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν αντιλαμβανόμαστε την ε, προστιθέμενη αξία, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα οποία δεν κοινοποιούνται στο κοινό πέραν του προγράμματος συστηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ορισμένες δραστηριότητες και με έντυπα και ε, με ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική εφημερίδα ε, και υπήρχε οπτικοακουστικό υλικό χωρίς όμως ε, να απαιτηθεί ε, να δίδονται λεπτομερείς ε, πληροφορίες οι οποίες δεν δίδονται στο κοινό και άρα όλα εξαρτώνται από την πρωτοβουλία των διαχειριστών του συγκεκριμένου προγράμματος ενώ θα μπορούσε κανείς να έχει αποκομίσει συμπεράσματα από τις βέλτιστες πρακτικές και από τις αποτυχίες όσον αφορά την αηφορία νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και την μακροχρόνια ε, διαχείριση των προγραμμάτων διότι εφόσον ε, αυτές ε, οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα μετά την αποπληρωμή του προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει πλέον πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά και βάσει αυτών των μειονεκτημάτων τα οποία έχουν εντοπιστεί θα καταλήξω τώρα στα σχόλιά μου και εις τις συστάσεις μου τα οποία θα εγγραφούν ή στο κείμενο για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν χαιρετίζω την έκθεση κατά δεύτερον λόγον ε, ε, σημειώνω ότι οι προσπάθειες συνέβαλαν τι ε, τις προσπάθειες διατηρήσεως των κρατών μελών και είναι υπέρ της διατήρησης των ειδών και ε, του χώρου τους, χώρου κατοικίας τους και ε, ε, υπήρξαν πολλές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη αλλά οι πόροι οι οποίοι αποδόθηκαν ε, απαιτούν να μπορέσει να υπάρχει καλή αξιοποίηση. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τον τρόπο επιλογής για να δώσει μία προτεραιότητα στις προτάσεις του LIFE και να ε, επιταχύνει τη διαδικασία επιλογής. Επίσης τονίζουμε ότι τα διαβήματα για την επιλογή δεν πρέπει να είναι πολύ μακροσκελή ε, για να μην υπονομεύσουν ε, τη διαδικασία αξιολόγησης. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις περιβαλλοντολογικές αρχές για να μπορέσει να καταρτήσει σωστά κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων όσον αφορά την αηφορία τους και τη βιωσιμότητά τους καθώς ε, αυτά τα θεσμικά όργανα έχουν εμπειρογνώμονες και μπορούν να προωθήσουν αυτά τα θέματα. Θα ζητούσα επίσης να αναλάβει προτεραιότητες για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της και να καταρτήσει ε, κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τη τη στρατηγική ενημέρωση ε, βάσει των ε, εμπειριών που έχει αποκομίσει και να δίδει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες έχει εντοπίσει. Θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συγχρηματοδότηση για μία ε, κατώτατη περίοδο παρακολούθησης αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και οι συμβατικές υποχρεώσεις θα πρέπει να προβλέπουν και τις ε, διαδικασίες ανάταξης θα πρέπει οι αρχές ε, της ε, συντηρήσεως της φύσεως να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά ε, μετά τη χρηματοδότηση τα προγράμματα του LIFE για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει βιωσιμότητα αφού ολοκληρωθεί η διάρκεια του προγράμματος να υπάρξουν σωστοί δείκτες επίσης για να αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος ήθελε ζήτησε το λόγο, δεν το βλέπω όμως πια έφυγε. Ο κύριος Σάλση από την Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να καλωσορίσω τις απόψεις ε, και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ελεκτικό συνέδριο θεώρησε ότι έχει βελτιωθεί το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την εισαγωγή του συστήματος LIFE το 1992. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία τώρα και να σας καταδείξω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις βασικές αρχές που ορίζονται στην έκθεση του Ελεκτικού συνεδρίου ότι το σχέδιο του LIFE οδηγεί στον ίδιο το σκοπό του προγράμματος γιατί γίνονται πολλές επενδύσεις ε, για πολλά χρόνια πολλές φορές και τα αποτελέσματα ο αντίκτυπος είναι ορατός μόλις μετά από εκατοντάδες χρόνια καμιά φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά το να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα θα έχουν το επιθυμητό αντίκτυπο στο τέλος της ε, δράσης τους και το γεγονός επίσης ότι τα προγράμματα αυτά εξακολουθούν να έχουν αξία προκειμένου να υπάρχουν αποτελέσματα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των οικοτόπων των ε, ειδών τα οποία έχει στο στόχο του το πρόγραμμα αυτό. Κάποια πρακτικά παραδείγματα πρόσφατων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ε, μας σύστησε το, Ευρωπαϊκό, το ελεγκτικό συνέδριο έχει γίνει, έχουμε πλέον δύο υπηρεσίες ε, στην μονάδα Life. Έχουμε την υπηρεσία Life, Life και Life Environment. Αυτό θα προλυάνει το δρόμο για την καλύτερη συγκέντρωση των δύο υπηρεσιών στους αντίστοιχους τομείς για τις οποίες είναι αρμόδιοι, αρμόδιες. Επίσης ξεκίνησε ε, μια ε, ανεπίσημη ε, διαδικασία διαβούλευσης. Ελπίζουμε να διαρκέσει αυτή η διαδικασία δύο-τρεις μήνες. Να είναι πολύ πιο σύντομη από ό,τι σήμερα δηλαδή και να χρησιμοποιηθούν και θέματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλες γενικές διευθύνσει, όπως τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας, για να εστιαστούμε, για παράδειγμα, στην πρόσθετη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για θέματα επικοινωνίας. Έχουμε βελτιώσει ήδη και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μας για να μεταδίδονται και να δημοσιεύονται όλα τα αποτελέσματα των διαφόρων προγραμμάτων. Επίσης, θέλουμε να θέσουμε σαφέστερες απαιτήσεις για τους δικαιούχους για να είμαστε σίγουροι ότι οι δικαιούχοι όταν μας υποβάλλουν ε, αναφορές ε, μας υποβάλλουν τα σωστά στοιχεία και επίσης εργαζόμαστε στο ότι αφορά τη δικτύωση. Δηλαδή διοργανώνουμε θεματικά σεμινάρια. Έγινε πρόσφατα ένα σεμινάριο για την Ιταλία και θέλουμε να υπάρχει μία διαδικασία, αν θέλετε, στα πλαίσια ενός δικτύου για την διανομή των αποτελεσμάτων. Ποιοι είναι σε θέση να διανέμουν τα αποτελέσματα για τα όσα μάθαμε και τα όσα διδαχτήκαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εξπόστο. Το 2002 δημοσίευσαμε ένα έργο, το Life After Life για την ε, σύνοψη και την επισκόπηση εννέα προγραμμάτων. Αυτό καταδεικνύει ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει το τι γίνεται μετά το πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και στο εγχειρίδιο αυτό είπαμε ότι σκοπός μας είναι να κοιτάξουμε ένα πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του. Και αυτό βάσει κριτηρίων ε, ποιοτικών και ποσοτικών σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να ομολογήσω ότι για να γίνει αυτό το μακροπρόθεσμο follow-up κάθε προγράμματος το οποίο έχουμε χρηματοδοτήσει μετά από χρόνια, μετά, από χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του αποτελεί ένα πραγματικά τεράστιο ε, έργο. Αυξήσαμε τις επισκέψεις ex post, για παράδειγμα, από 10 σε 15%. Αυτό καταδεικνύει ότι επενδύουμε όσο μπορούμε στον τομέα αυτό. Συνολικά, συμφωνούμε ουσιαστικά με όλες τις ε, συστάσεις της έκθεσης και προφανώς και με τον τρόπο που τα παρουσίασε όλα αυτά η συγκήτρια του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ένα στοιχείο μας απασχολεί. Το να μπουν συμβατικές υποχρεώσεις ε, στην συμφωνία για να διατηρηθούν για μια περίοδο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε από συμβατική άποψη για να επιβάλλουμε νομικές υποχρεώσεις και κάποια από τα στοιχεία αυτά αποτελούν τμήματα της ε, πρακτικής φύσεως. για παράδειγμα θέματα αγορών. Έχουμε επίσης ε, ε, πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τα βιώσιμα αγαθά, όπως οι υποδομές, για 10 χρόνια συνήθως. Πολύ προσοχή δίνουμε και για τα διαχειριστικά σχέδια, προκειμένου να ε, εγκρίνονται νομοθετικά, νομικά πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, αυτό αποτέλεσε πρόβλημα. Αυτό που θα πρέπει να οριστεί ακόμα από σημαντική άποψη είναι το θέμα του προσωπικού. Τι χρειάζεται δηλαδή ο δικαιούχος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί ο αντικτύπος του, προγράμμα, του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του προσωπικό. Και αυτό λοιπόν το εξετάσαμε και με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι νομικά και πρακτικά αδύνατον να τεθούν τέτοιες κυρώσεις από νομικής άποψης. Θεωρούμε ότι μια θετική προσέγγιση, όπως αναφέρεται στην πρώτη σύσταση του Ελεκτικού Συνεδρίου, να δοθεί δηλαδή προτεραιότητα σε κάποια προγράμματα τα οποία φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο βαθμό ε, βιωσιμότητα κατά τη φάση της επιλογής, πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί ένα σωστό μέτρο και θα πρέπει να βελτιωθεί η μέθοδος αυτή. Και τέλος, να αναφέρω ότι η δική μας εμπειρία και από αυτό φαίνεται και από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου φαίνεται ότι στην πραγματικότητα τα προγράμματα τα οποία τα εγκαταλείπουμε μετά την ολοκλήρωσή του στα πλαίσια του LIFE, είναι ουσιαστικά μηδαμινά. Δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Και βλέπουμε ότι τα προγράμματά μας έχουν αντίκτυπο. Συμβάλλουν στην προστασία της φύσης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκαϊέρ. Καταρχήν, ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καζαμία και τους ε, συναδέλφους τους, καθώς επίσης και την κυρία Ιβάνοβα για το έγγραφο εργασίας διότι πιστεύω ότι όλα τα θέματα όπου υπάρχουν ελλείψεις αναφέρθηκαν. Έχω όμως δύο ερωτήσεις που ε, θέλω να απευθύνω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μία είναι σχετικά με την διατύπωση εις το ελεγκτικό, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι μειώθηκαν ε, οι ε, οι διαφορές και ότι το πρόγραμμα LIFE ε, αξιολογήθηκε με ίσα κριτήρια και πιο δίκαια κριτήρια. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, στο θέμα της αξιολόγησης περιορίστηκε το, η αξιολόγηση μόνο στην βιωσιμότητα. Όταν βλέπω όμως τον πίνακα του ελεκτικού συνεδρίου βλέπω ότι ποσοστιαία η βιωσιμότητα έχει σχεδόν εξαφανιστεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Και μετά διαβάζω σε ένα άλλο σημείο ότι οι πληροφορίες ε, τις οποίες μπορούμε να αποκομίσουμε επίσης ε, παρουσιάζουν ελλείψεις ε, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο γίνεται με τα χρήματα των φορολογιουμένων στα προγράμματα LIFE και τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουμε δεν ε, αποδεικνύουν επαρκώς την αποδοτικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι στο ότι 15% των προγραμμάτων θα μπορούσαν να έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το τέλος της εφαρμογής τους και θα ήθελα να ξέρω αν χρειάζεται να διευρυνθεί και κατά πόσον ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος για να μπορέσει να υπάρξει μια εκ των υστέρων αξιολόγηση κατά 100% δηλαδή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, νομίζω ότι είδαμε ένα από τα μέτρα τα οποία ήταν πολύ αμφιλεγόμενα τουλάχιστον σε μία χώρα να επιληθεί ε, ειρηνικά. Βλέπω ότι όλα τα θέματα για το 2004 τουλάχιστον ε, έχουν επιληθεί, υπήρχε σωστή χρηματοδότηση και όλα αυτά συνέβαλαν πολύ ε, στο να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Όσον αφορά το πρόγραμμα προστασίας των πουλιών και ε, μετά από αυτά τα οποία ο κύριος Γκάγερ ήθελα να ρωτήσω πώς υπολογίζεται ότι θα είναι οι ανάγκες του προγράμματος για τα επόμενα έτη διότι πιστεύω ότι μάλλον θα διονγκωθούν παλά θα περιοριστούν. Κυρία Ματή, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ είμαι σαν τους, ε, σκέφτομαι σαν τους συναδέλφους. όλοι τρέφαμε ελπίδες για αυτές τις πιστώσεις, διότι οι πολίτες ε, μιλούν πολύ για όλα αυτά τα ποσά και στην προεκλογική εκστρατεία ήταν και ένα μπούμεραγκ διότι μιλάμε πολύ για περιβάλλον αλλά όταν οι ευρωσκεπτικιστές λένε ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε εδώ ένα εργοστάσιο λόγω ενός ε, μιας ράτσας καραβαίων ή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο έργο λόγω μιας πεταλούδας ε, ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα πολλές φορές. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν Ε, ποια είναι η πραγματική επίπτωση της επιστροφής αυτών των γεών, ε, πώς, ε, ποια είναι η επίπτωση στη χλωρίδα και στην πανίδα. Διότι φυσικά όλοι θέλουμε Ε, το καλό του πλανήτη αλλά όταν κόβουμε τη χρηματοδότηση για αυτές τις περιοχές ε, πραγματικά ε, σπαταλούμε τα χρήματα του φορολογούμενου. Ο κύριος Σάλση για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω με τη σειρά που τέθηκαν τα ερωτήματα. Τα κριτήρια βιωσιμότητας μειώθηκαν ως προς τον αντίκτυπο και το τον αριθμό των προγραμμάτων. Επειδή η διαδικασία επιλογής ε, συμπυκνώθηκε σε μία διαδικασία όπου μία υπηρεσία πλέον διαχειρίζεται το πρόγραμμα live με ένα πρόγραμμα αξιολόγησης των προγραμμάτων. Σας διαβεβαιώ ωστόσο ότι θα υπάρξει μία αναθεώρηση, ίσως όχι στην παρούσα φάση, γιατί έχουν δημοσιευτεί τα κριτήρια επιλογής και θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουν δημοσιευτεί. Όχι λοιπόν για τα εφιστάμενα προγράμματα, αλλά για τον επόμενο γύρο. Ιδιαίτερα εφόσον αλλάζουμε τον τρόπο υποβολής των προγραμμάτων επιλογής και ε, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα θέματα τώρα για νομής. Φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής οι δράσεις μας. Από τότε που ξεκίνησα στο live το 1994, θυμάμαι και μια απόφαση του 1995 που ανέφερα ότι εδώ δεν είναι επαρκής η δράση μας. Αυτό αληθεύει εν μέρη, αλλά εν μέρη δεν αληθεύει κιόλα. Γιατί εμείς ως Επιτροπή καταβάλαμε μια σημαντική προσπάθεια στον τομέα αυτό για την ε, διάδοση ουσιαστικά των πληροφοριών και των στοιχείων στα πλαίσια του LIFE. Αλλά εκ παραλλήλου συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά πολλά από τα στοιχεία αυτά. Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο, καλύτερη ιστοσελίδα, να διοργανώνουμε πιο πολλά εργαστήρια για να βελτιώσουμε αυτά τα θέματα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να περάσουμε από την απλή διάδοση των στοιχείων ουσιαστικά στην ουσιαστική επικοινωνία. Προκειμένου να στέλνουμε τις πληροφορίες αυτές στα κατάλληλα άτομα. Και γι' αυτό λοιπόν ε, επενδύουμε τώρα σε αυτή την πολυτομιακή, αν θέλετε, ε, μετάδοση των πληροφοριών, σεμινάρια, εργαστήρια, όπου συναντιούνται οι εμπειρογνώμονες και συζητούν τα θέματα τα οποία αυτά γνωρίζουν. Και νομίζουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική συμβολή του θέματος αυτού. Σε ό,τι αφορά την ε, ex post παρακολούθηση των προγραμμάτων, 15% πλέον είναι το ποσοστό Στην πραγματικότητα το 15% αυτό αποτελεί μόνο ένα τμήμα των όσων κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά έχουμε σε πολλές περιπτώσεις ε, μία αναφορά από τους ίδιους τους δικαιούχους και αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθάμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Και εγώ εκτιμώ ότι το πραγματικό ποσοστό παρακολούθησης εξπόστων των προγραμμάτων είναι γύρω στο 50%. Όλα τα προγράμματα δέχονται τουλάχιστον μία επίσκεψη με την, μετά την ολοκλήρωσή τους. Και επίσης μία ερώτηση που τέθηκε για το επίπεδο ζήτησης. Θα περιμέναμε ότι θα είχε αυξηθεί το επίπεδο αυτό. Αλλά δυστυχώς, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η οικονομική κρίση χτύπησε τον τομέα αυτό όπως και πολλούς άλλους και έχει μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων τα τελευταία τρία χρόνια και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το life nature. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα δημόσια ταμεία. Και όταν οι δημόσιες ε, οι δημόσιοι αυτοί πόροι ε, δεν είναι πλέον ε, άφθονοι. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τα κράτη-μέλη να βρουν τη χρηματοδότηση αυτή. Αν θέλουμε λοιπόν σήμερα να λειτουργήσει καλύτερα το Life Nature, θα πρέπει να διαμορφωθεί με πιο ευέλικτο τρόπο και όχι με πιο αυστηρό σημαντικό τρόπο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν. Και η ίδια η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα δεν αμφισβητείται γιατί εν γέννη πρόκειται για βιώσιμα προγράμματα. Κάποιες δράσεις εντός ορισμένων προγραμμάτων μπορεί να μην είναι τόσο βιώσιμες, αλλά σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να σας μιλήσω επάπειρον για την βιωσιμότητα του Life Nature, αλλά να σας ε, δώσω κάποια σύντομα παραδείγματα. Το 1995, σε μια οδηγία στο άρθρο 6, αναφέρθηκε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν τα, τις τοποθεσίες Natura 2000. Πέντε εξ αυτών ε, χρηματοδοτήθηκαν Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Η Ιταλία ήταν η πρώτη που το 1995 υπέβαλε κατάλογο ως αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού. Και αναπτύσσουμε τον κατάλογο αυτό από το 1995. Θεωρώ για ένα τόσο μικρό πρόγραμμα όπως το Life Nature να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην πολιτική είναι πραγματικά ένιγμα το πώς το πετύχαμε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα για τον συνάδελφο από τον Ακτικό Συνέδριο είναι η ίδια η Ελλάδα. Η Ελλάδα το 1992 δεν είχε ουσιαστικά μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίε θα μπορούσαν να, ε, να εκτελέσουν τέτοια προγράμματα διατήρησης ε, τη φυση Είχαν σεμινάρια, εργαστήρια, όχι όχι τέτοια προγράμματα του ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Και μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν αρκετέ μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Ελλάδα που είναι με το παραπάνω ικανέ να εκτελέσουν τέτοια προγράμματα. Μιλάμε λοιπόν για ανάπτυξη δυναμικού, η οποία είναι βιώσιμη, πιστέψτε με. Grazie. Λοιπόν, σα θυμίζω, η επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα είναι 10 Νοεμβρίου, όπου θα παρουσιάσουμε και την ετήσια έκθεση 2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεδριάζουμε επίση 2 Δεκεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου. Στι 12.30 θα φύγει το λεωφορείο για να επισκεφθούμε το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα θα διέκοπτα μισή ώρα για να συνεχίσουμε στις 12 διότι ξέρω ότι συνεδριάζουν οι διάφοροι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων και θα έχουν αποφασίσει μέχρι τις 12. Η γραμματεία πάντως μας έχει δώσει εδώ ένα πρόχειρο το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε για αυτά τα πέντε σημεία. Στις 12 ξανασυνεδριάζουμε λοιπόν για πέντε λεπτά.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 Siamo solo io e lei. Allora io direi di eh, giusto prendere un attimo. Λοιπόν, εγώ λέω να σας πω το εξή και μετά να φεύγουμε. Μου είπανε ότι στις συνεδρίες των ομάδων για, τις, για το κατάλογο των προτεραιοτήτων Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τον κατάλογό της που εμείς τον έχουμε. Άλντε, Έλκε και Σοσιαλιστές. Δύο κοινά σημεία μου έχουν επισημάνει. τον δημοσιονομικό κανονισμό, την βελτίωσή του και το περιθώριο λάθους που μπορεί να υπάρχει. Επίσης, υπάρχουν κοινά σημεία για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, την Όλαφ, απλούστευση δημοσιονομικού κανονισμού, δημοσίευση των ονομάτων των δικαιούχων κλπ. Τώρα πρέπει να φεύγουμε γιατί 12.30 πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο. Τώρα για το ελεγκτικό συνέδριο θα δώσουμε και τον κατάλογο μετά εκεί των ομάδων μία προς μία. Ευχαριστώ.